Καλημέρα σα, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είστε πολλοί, κάποιοι τέλο πάντων. Καταρχάς να σα πω ότι δεν θα υπάρχει διερμηνία από τα ρουμανικά, από και προ τα ρουμανικά. Αλλά σήμερα το πρωί μόνο. Δεν θα υπάρχει δηλαδή η ρουμανική, δεν θα υπάρχουν διερμηνείς ε, στην ρουμανική καμπίνα. διότι έχουμε διερμηνείς που είναι άρρωστοι. Τώρα το απόγευμα μπορεί να αναρρώσουν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων, θα ήθελα ε, λέει η εκπρόσωπος από την ε, Ρουμανία ότι ε, θα ήθελα να σημειώσετε ότι θέλουμε πάντα καμπίνα, ρουμανική καμπίνα και στην Επιτροπή μας και στην, στις υποεπιτροπές στην ομάδα εργασίας. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ζητήσω να φροντίσετε να βρούμε, να υπάρχει πάντα διερμηνία. Καλώς, ε, λέει ο Πρόεδρος, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ε, και εγώ θεωρώ ότι καλό θα είναι να έχουμε ε, διερμηνείς. Η γραμματεία όμως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, διότι ξέρουν ότι και μένα με ενδιαφέρει, θέλουμε όλες οι καμπίνες να εκπροσωπούνται εδώ. Αλλά κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα να το τονίσω αυτός, στα τρία-τέσσερα άτομα τα οποία είναι παρόντα στην αίθουσα και ξέρω ότι δεν, ε, τα, δεν πρέπει να τα λέω σε εσά, πρέπει να τα λέω σε όλου του υπόλοιπου, αλλά οι διερμηνεί είναι περισσότεροι από ότι οι βουλευτέ. Λοιπόν, να μαζεύουμε όλου αυτού του διερμηνεί και να μην υπάρχουν ε, βουλευτέ στην αίθουσα, τι να σα πω, αυτό έχει αρχίσει και με εκνευρίζει λιγάκι. Πραγματικά ε, τι να σας πω, είμαστε, πληρωνόμαστε όλοι για να συμμετέχουμε στις ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής και είμαστε απόντες. Ζητάμε πάντα να υπάρχει διερμηνία για όλες τις γλώσσες, αλλά εφόσον ζητάμε διερμηνία, τουλάχιστον να έχουμε και, και συναδέλφους. Δεν έχει σημασία αν είναι μεγάλες ή μικρές γλώσσες, μεγάλες ή μικρές χώρες. Ε, πρέπει να έχουμε όλη την δυνατότητα να ακούμε ε, τις παρεμβάσεις στη γλώσσα μας. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, ας επανέλθουμε στα θέματά μας, ε, έχουμε ε, εκπροσώπους της Κομισιό μαζί μας. Έχουμε την κυρία Στέφανη Μίτσελ, που είναι υπεύθυνη για τα θέματα που μας, θα μας απασχολήσουν σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τις τρεις ε, εκπροσώπους Γενικής Διεύθυνσης που ήρθατε εδώ σήμερα μαζί μας, γιατί δείχνει ακριβώς ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα ε, για την Επιτροπή μας. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί νέοι από την Ευρώπη ε, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αποφασίσαμε να δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες ε, τι ακριβώς συμβαίνει και τελικά όμως μάθαμε, ψάχνοντας, ε, είδαμε ότι η Κομισιόν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν το ξέραμε, γιατί δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε όλα, δεν μπορούμε να ενημερωνόμαστε για τα πάντα, αλλά ε, πιστεύω ότι επειδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, ε, θα ήθελα όλοι να τα ακούσουμε αυτά. Βέβαια όλοι δεν είναι εδώ, αλλά δεν έχει σημασία, έστω και αυτοί οι happy few τέλος πάντων, να ενημερωθούμε γιατί πρόκειται για θέματα τα οποία είναι σημαντικά για το μέλλον της Ευρώπης. Το αν έχουμε αρκετές επιχειρήσεις, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ε, χρεοκοπήσουν αυτές ε, οι, οι επιχειρήσεις ή εάν αναγκαστούν να κηρύξουν πτώχευση, πώς αυτό μπορεί να γίνει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι σημαντικά και ε, καλό θα είναι να ακούσουμε την Κομισιό, να μας πει τι έχει κάνει, ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε και αν θέλετε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ε, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις. Στις 10, ε, μέχρι τις 10 έχουμε την, ε, την δυνατότητα να συζητήσουμε γιατί στις 10 ξεκινάνε οι ψηφοφορίες. Να είσαστε σίγουροι ότι τότε θα γεμίσει η, η, η αίθουσα. Τέλος πάντων ας ξεκινήσουμε με την Κομισιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. πριν από μερικά χρόνια ο Γενικό Διευθυντής μα, όταν συζητούσαμε πώ κάποια project συνδέονται με κάποια άλλα και ποιε είναι οι δυσκολίε συντονισμού είπε ότι αν ήξερε η Κομισιόν, τι ξέρει η Κομισιόν, θα γινόντουσαν πολλά πράγματα. Τώρα όμω η Κομισιόν γνωρίζει αρκετά πράγματα και καλό θα είναι να, και εσείς και εμείς να ξέρουμε τι ξέρουμε, ε, γιατί όντως όλοι μαζί ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα για λίγα λεπτά να σας ε, πω τι έχουμε κάνει σε αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα και μετά η συνάδελφός μου θα προσθέσει κάποια πράγματα και μετά θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο περιβάλλεται, αν θέλετε, και από άλλα συμπληρωματικά θέματα. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις. Ξέρετε ότι τουλάχιστον το 50% των επιχειρήσεων επιβιώνουν τα επόμενα 5 χρόνια από την στιγμή που δημιουργούνται και το 15% των επιχειρήσεων που κλείνουν οφείλονται στη πτώχευση. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε όμως είναι ότι μόνο 4 έως 6% των πτωχεύσεων είναι, ε, συνδέονται με κάποια απάτη, με κάποια, ε, κάποια δικήματα ή κάποια συμπεριφορά παράνομη. Δόλια συμπεριφορά. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν χρειάζεται, δεν τα ξέρει το γενικότερο κοινό, δεν τα ξέρει ούτως ή άλλως και ο επιχειρηματικός κόσμος. Εάν ρωτήσουμε τι φοβάται ο κόσμος και δεν δημιουργεί μία επιχείρηση, ο πρώτος κίνδυνος τον οποίο αναφέρουν είναι ο κίνδυνος πτώχευσης. Η δεύτερη απάντηση είναι η αβεβαιότητα των εσόδων. Και το, ο τρίτος είναι ότι θα πρέπει να χάσουν όλα του τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή τα πάντα. Και ναι, μεν οι επιχειρηματίες ε, αρέσκονται στον κίνδυνο, αλλά και ο κίνδυνος να χάσουν τα πάντα ε, είναι πολύ μεγάλος για να προχωρήσουν. έχουμε δύο συνέπειες. Έχουμε την συνέπ, τις άμεσες συνέπειες σε αυτούς που είναι ήδη επιχειρηματίες, σε αυτούς που έχουν κάνει ήδη τη βουτιά τέλος πάντων και που αντι, αντιμετωπίζουν κάποιες, ε, κάποιους κινδύνους από, και από το νομικό πλαίσιο ε, και που αισθάνονται αποθαρρυμένοι, δεν θέλουν να προχωρήσουν, δεν θέλουν να διευρύνουν τις επιχειρήσεις τους ε, και δεν είναι μόνο το ψυχολογικό στοιχείο αλλά είναι και πρακτική αδυναμία ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες επομένως ε, ε, ίσως πρακτικά, να είναι πρακτικά αδύνατο να ξεκινήσουν ξανά στο 95-96% θεωρείται αδύνατον τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση να είναι, ε, να είναι ή να είναι ανέντιμοι κτλ. Στην μεγάλη πλειοψηφία των πτωχεύσεων, των χροκοπιών, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα, μια σειρά ε, γεγονότων τα οποία ενεργοποιούνται από κάποιο λογαριασμό ο οποίος δεν πληρώθηκε κάποιος πελάτη που δεν πλήρωσε κάποια προμήθεια που δεν έγινε και υπάρχει μια σειρά τυχών γεγονότων ενδεχόμενα και λόγω μια μικρή ανικανότητας να διαχειριστούν την κατάσταση, όχι όμως λόγω ε, παρανομίας ή δόλια συμπεριφοράς. Τώρα μια επιχείρηση που ξεκινάει ε, δεύτερη φορά μπορεί να έχει, μια, να έχει μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, να μπορεί να διευρυνθεί περισσότερο. Υπάρχει τώρα και μια άλλη μια συνέπεια που είναι είναι, είναι ε, οι επιχειρηματίες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδυνάμοι επιχειρηματίες αλλά που δεν ξεκινάνε ποτέ διότι ακριβώς ξεκινάνε με μια σειρά προβλημάτων. Δείτε κάποιους δείκτες του ευρωμαρομέτρου. Από το 2009 είδαμε μόνο ότι το 45% των Ευρωπαίων θα θέλανε να είναι αυτοαπασχολούμενοι ε, και και θα ήθελαν να είναι υπάλληλοι. Ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείε η κατάσταση είναι ακριβώ το αντίθετο. Εάν ε, συγκριθούμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε ή με την Ασία ενδεχόμενα, υπάρχει ένα επιχειρηματικό χάσμα, υπάρχει ένα κενό και εκεί θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Εάν στο ευρωμαρόμετρο, ευρωμαρόμετρο ε, αφήναμε τη δυνατότητα να σχολιάσουν τα άτομα με, τις, με κάποιες δηλώσεις, ε, η, δήλωση που θα έκανε ήταν ότι στο, ερώτημα δεν ξεκινάω μια επιχείρηση γιατί θεωρώ ότι θα χρεοκοπήσω. Το 48% των Ευρωπαίων απήντησαν ότι ναι, όντως αυτός είναι ένα υπαρκτός φόβος. Ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείε αυτό δεν υπάρχει. Μέχρι τώρα Υπάρχουν δύο νομοθετήματα, 1346-2000 ε, που είναι ε, τη διαδικασία πτώχευσης και ασχολείται με την ε, δικαιοδοσία που είναι υπεύθυνη όταν το θέμα είναι διασυνοριακό και την αναγνώριση των αποφάσεων των δικαστικών διασυνοριακό και το νομοθέτημα που προστατεύει τους εργαζόμενους. Και θα έλεγα ότι ο στόχος είναι να υπάρχει ισότητα δικαιωμάτων για όλους ε, σε περίπτωση διασυνοριακών υποθέσεων ενδοκινοτικών και ως προς την διαδικασία. Η διαδικασία βρίσκεται στην αρχή ε, και θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και ε, ε, μόλις αρχίζει η διαδικασία, ε, πυροδοτείται μόλις υπάρχει η πτώχευση. Εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε πόσο μπορούμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες. Μελέτες του 2004, του 2005 ασχολήθηκαν με το θέμα και το 2007 μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να υπερνικήσουμε το στίγμα αυτό της αποτυχίας της επιχειρηματικής ένα σύστημα σε ολόκληρο την Ευρώπη. Το 2008 στην πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να προωθήσουν μια θετική στάση ούτως ώστε να δώσουν στους νέους επιχειρηματίες μια νέα εκκίνηση. Επίσης ασχοληθήκαμε με τα start-ups, τις νέες μικρές επιχειρήσεις για να τις υποστηρίξουμε και τελικά και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την σημερινή μας συζήτηση, ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να καταστήσουν εφικτό όλες οι νομικές διαδικασίες για την εκαθάριση των επιχειρήσεων σε περίπτωση μη δολίας πτώχευσης να μπορούν να περατώνονται μέσα σε ένα χρόνο. Βεβαίως ε, είναι ο ευκολότερος δρόμος αλλά και ο σκληρότερος, ο πιο δύσκολος. Η μέση διάρκεια στις, ε, στα 27 κράτη-μέλη για την εκαθάριση μιας επιχείρησης ε, είναι λίγο κάτω από δύο χρόνια στην Ιρλανδία, σε τέσσερα δέκατα του χρόνου στην Σλοβακία χρειάζονται τέσσερα χρόνια για την εκαθάριση. Όλες οι άλλες χώρες είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Εξετάσαμε λοιπόν την, τον, τον νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να προωθήσουν τη δεύτερη ευκαιρία για μικρούς επιχειρηματίες περιορίζοντας την διάρκεια για την εκαθάριση των ε, χρεών. Ε, να έχουμε τρία χρόνια στο ε, περισσότερο. Ένα χρόνο για εκαθάριση και τρία χρόνια κατά τις οποίες οι οφειλέτες μπορούν ε, να κινούνται. Έχουμε μια πύλη ε, στην που δίνει ε, πληροφορίες για τα θέματα αυτά και έχουμε επίσης ένα ολόκληρο φάσμα γνώσεων και πληροφοριών και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο για να σας μιλήσει για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Η πτώχευση αυτή καθεαυτή ως λέξη είναι πάρα πολύ άσχημη λέξη. Πολύ δυσάρεστη και είναι, είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας όπου υπάρχουν αντιδράσεις από παντού μόλις αναφέρεται αυτή η λέξη. Είναι λοιπόν ένα, δεύτερο θέμα, ένα δύσκολο θέμα για να ασχοληθεί κανείς με αυτό. Κανείς δεν φαίνεται πρόθυμος να μιλήσει για αυτή την πτώχευση. Μιλάμε για αποτυχία. Γιατί εξετάσαμε το θέμα αυτό από την άποψη της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων. Η πτώχευση και η δεύτερη ευκαιρία και είναι μια διαδικασία, κυρίως η δεύτερη ευκαιρία, η ροή αυτή. Η πτώχευση δεν συμβαίνει γιατί κάποια μέρα ξυπνάτε και συμβαίνει αυτό. Είναι μια ολόκληρη ροή. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να έχουν ε, να έχουν προβλήματα, αρχίζουν τυπική άτυπη αναδιάρθρωση, μπορεί να έχουν πτώχευση, μπορεί ε, να μην πτωχεύσουν, μπορεί να γίνει κάποια στάση πληρωμών. Σε αυτήν την γραμμή των γεγονότων, αυτό που κάναμε με την πάροδο των ετών, και αρχίσαμε στη δεκαετία του 90 είναι να αναλύσουμε από την άποψη του επιχειρηματίου ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις της πτώχευσης και της δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό το οποίο είδαμε εδώ ότι υπάρχει, ε, υπάρχουν δυνατότητες, μαζικές δυνατότητες ε, μέτρων και δυνατοτήτων ε, που δεν λήφθηκαν υπόψη από τις αρχές. Μπορούμε να αναφερθούμε στην προσωπική αφαιρεγγιότητα, διότι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε εδώ είναι να συγκεντρωθούμε ε, στην δεύτερη ευκαιρία, να δώσουμε ένα σήμα στους επιχειρηματίες ότι θα υπάρξει μια δεύτερη ευκαιρία. Ότι η επιχειρηματικότητα ε, δεν είναι μια ισόβια καταδίκη. Ότι μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Το σημαντικό λοιπόν είναι να εστιαστούμε στην προσωπική αφαιρεγγιότητα. Όταν μια εταιρεία πεθαίνει, πεθαίνει, δεν συμβαίνει τίποτα. Τι γίνεται με τον επιχειρηματία όταν πτωχεύει, τι συμβαίνει τότε. Η Στεφανία ανέφερε δύο σημαντικά πράγματα. Είναι ότι ο τομέας αυτό το θέμα αυτό δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά από τις αρχές. Υπάρχουν δύο επιπτώσεις σοβαρές. Έχουμε επιχειρηματίες που έχουν πτωχεύσει, που είναι επιχειρηματίες και δεν Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να έχουμε τώρα επιχειρηματίες στην Ευρώπη, να έχουν το πνεύμα το επιχειρηματικό σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες, έχουν την πείρα του management, μαθαίνουν από την πείρα τους και θα γίνουν καλύτεροι τη δεύτερη φορά, θα βελτιωθούν, αλλά όχι μόνο αυτό. Οι συνέπειες είναι ακόμα μεγαλύτερες και όπως είπε η Στεφανή, υπάρχει μια διάχυση σε όλο το σώμα, τον κόσμο των επιχειρηματιών. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι ε, και δεν έχουμε πια τόσους πολλούς νέους στην Ευρώπη. Πολλοί νέοι στην Ευρώπη δεν αρχίζουν την εταιρεία τους διότι φοβούνται μήπως αποτύχουν. Ας δούμε μια από τις τελευταίες μελέτες για το θέμα που είναι το ευρωβαρόμετρο σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Κατά μέσο όρο στην Ευρώπη 50% του πληθυσμού συμφωνεί με το γεγονός ότι κάποιος δεν πρέπει να αρχίσει μια επιχείρηση αν υπάρχει κίνδυνος να αποτύχει η επιχείρηση και ο κίνδυνος είναι κάπως ταυτόσημα και έχουμε εδώ ένα μήνυμα πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν 50% που φοβούνται να αρχίσουν μια επιχείρηση διότι φοβούνται ότι θα αποτύχουν, θα πτωχεύσουν. Αυτό το ποσοστό δεν είναι ενθαρρυντικό. Αν συγκρίνουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες, ο αριθμός είναι 26%. Είμαστε λοιπόν πολύ χειρότεροι, διπλά χειρότεροι από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και έχουμε επίσης στην Κίνα 23%. Δεν είναι μόνο λοιπόν η Αμερική, είναι και η Κίνα, οι δύο βασικοί μας ανταγωνιστές παγκοσμίω έχουν μια στάση με μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα. Είναι έτοιμοι να αναλάβουν τον κίνδυνο να ανοίξουν μια επιχείρηση πολύ περισσότερη από ό,τι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν χάνει ένα μεγάλο κεφάλαιο επιχειρηματικότητας λόγω της κατάστασης αυτής και της στάσης που έχουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο σε τομείς που μας ενδιαφέρουν, η προχωρημένη τεχνολογία όπου έχουμε ε, επιχειρηματίες και επιστήμονες που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα. Είναι άνθρωποι που έχουν επιλογή, που πηγαίνουν να εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ερευνητικά κέντρα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν την επιλογή και δεν θέλουν να αναλάβουν τον κίνδυνο. Νομίζω λοιπόν ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι εμείς ως Ευρωπαίοι χάνουμε μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. Όχι μόνο για τους επιχειρηματίες οι οποίοι πτωχεύουν, αλλά τους επιχειρηματίες που δεν θέλουν καν να ανοίξουν μια επιχείρηση. Έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων βάσει της σύσταση και έχουμε εμπειρογνώμονε από Υπουργεία από τα 27 κράτη-μέλη και άλλων χωρών, δηλαδή 33 χώρες εκπροσωπούνται σε αυτή την ομάδα και παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία την πτωχευτική για να βοηθήσουμε ε, τους ε, επιχειρηματίες ε, να ξαναρχίσουν. Ε, να... Είναι ένα έγγραφο το οποίο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο που ανέφερε η Στέφανη. Είναι 12 σελίδες με μερικές ενδείξεις του τι μπορεί να κάνει για να προλάβει την πτώχευση, την νομική διαδικασία, την δικαστική διαδικασία και να έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Έχουμε τα διάφορα βήματα τα διάφορα στάδια. Ένα πράγμα το οποίο διαπιστώσαμε και αυτό δεν μας εκπλήσει ως ένα βαθμό, όταν πτωχεύει μια επιχείρηση, όταν αρχίζει η διαδικασία, είναι ήδη πάρα πολύ αργά. Όταν μιλάμε λοιπόν για πτώχευση, δεν θα πρέπει να μιλάμε για την ίδια την πτώχευση, να εστιαζόμαστε στη νομική διαδικασία την πτωχευτική, αλλά στην πρόληψη της πτώχευσης. Τι μπορούμε να κάνουμε πριν για να βεβαιωθούμε ότι το κεφάλαιο το ανθρώπινο και οικονομικό να μην χαθεί και όταν ε, η εταιρεία και κυρίως ο επιχειρηματίας πτωχεύσει, πώς μπορούμε να ανακτήσουμε αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο για να επιτρέψουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερη ανάπτυξη. Η σημαντικότερη σύσταση του SBA είναι ότι ε, προτείνουμε ή ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να υπάρχει ε, πλήρης απαλλαγή σε περίοδο τριετή ε, μετά να κλείσει η διαδικασία ε, της υπτωχευτική και να δώσουμε στον επιχειρηματία για να είναι ελεύθερος χρεών και να μπορεί να ξαναρχίσει μια νέα εταιρεία. Πάρα πολλές μελέτες επιβεβαιώνουν αυτήν την σύσταση η οποία δεν ήρθε από το πουθενά. Το Insol Service επίσης έκανε μια μελέτη το 2001 όπου μας λέει ότι η διάρκεια δεν θα έπρεπε να ξεπερνάει τα τέσσερα χρόνια και θα έπρεπε κατά προτίμηση να είναι τριετής. Αυτή είναι μια διεθνής μελέτη που έγινε από έναν εξάρτητο σώμα. Επίσης έγιναν άλλες μελέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιμένουν πάνω στο γεγονός ότι η διάρκεια θα πρέπει να είναι στο maximum τρίτης Το 2006 ο Ολλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης οργάνωσε ένα σεμινάριο και κάλεσε Δανούς, Γάλλους, Λετωνούς, Λουξεμβούριους και Σουηδούς από τις αρχές δείχνοντας ότι το σύστημά τους διεκπεραιώνεται σε λιγότερο από τρία χρόνια και οι αρχές συμφωνούν. Αυτή η απαλλαγή απαιτείται ε, και όταν τα κράτη θέτουν αυτήν την διάρκεια θα πρέπει να είναι maximum τριετής η διάρκεια. Υπάρχουν ε, βεβαίως μερικές αποδείξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου εκεί χρειάζεται μόνο ένα έτος σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από τρεις ή έξι μήνες ε, δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης ε, περαιτέρω ε, χρεών, οφειλών. Και για τους πιστωτές το γεγονός ότι κρατάτε το ένα άτομο έτσι ενεωρήσει δεν οδηγεί σε κανένα οικονομικό όφελος, ενώ παρεμποδίζεται η επανεκκίνηση μιας νέας εταιρείας η οποία σε μικρό ή μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να ανακτήσει τις απώλειες της πρώτης υπόθεσης. Έχουμε και άλλες πληροφορίες για όλα αυτά τα στοιχεία. Βεβαίως περιλαμβάνονται όλα και στην ιστοσελίδα μας και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι πρέπει όντως να πάρουμε κάποια μέτρα για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους επιχειρηματίες, ειδικά σήμερα, σε αυτή την κατάσταση έτσι όπως έχει, ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι καταδίκη, ισόβια, και βεβαίως ε, δεν θα έχετε δεύτερη ευκαιρία δεν, και ότι δεν είναι καταδικαστικό αν κάποιος έχει μια αποτυχία. Όλοι έχουμε αποτύχει στη ζωή, αλλά φανταστείτε πώς είναι μια κατάσταση όταν κάνει κάποιος ε, ένα λάθος και τελειώνει. Μετά δεν έχει καμία δεύτερη ευκαιρία. Δεν μπορούμε λοιπόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον να κάνουμε κάτι τέτοιο και νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς την ύπαρξη, τη δημιουργία μιας δεύτερης ευκαιρίας για τους επιχειρηματίες. Ένα λεπτό. Θα ήθελα μια παρατήρηση να κάνω, γιατί χτες σύντομα το κάναμε και θα ήθελα να το ξανακάνω σήμερα. Έχουμε 20 δασκάλους μαζί μας από τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό New Energy για το έξιμο πρόγραμμα, για, την, για το πρόγραμμα για την ευφυή e e ενεργεία, ενέργεια. Ε, μαθητές λοιπόν που ε, με τους καθηγητές τους βεβαίως που κέρδισαν στον διαγωνισμό αυτό σήμερα είναι μαζί μας εδώ. Καλώς ήρθατε, τους ε, χαίρομαι πολύ που είσαστε μαζί μας. Ε, κάθονται εκεί πίσω και τους ξέχασα πιο πριν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα, παρακαλώ. Ήθελα απλώς να, πω, να κάνω ένα σχόλιο πριν από τέσσερις εβδομάδες Ολοκληρώσαμε μία προετοιμασία για ένα φυλάδιο που προετοιμάζουμε κάθε, ε, κάθε χρόνο με την, ε, το μυστικό της επιτυχίας. Ε, το έχουμε γράψει σε όλες τις γλώσσες. Έχουμε κάποια δείγματα και για τα μέλη της Επιτροπής σας. Αν θέλετε περισσότερα δείγματα στην γλώσσα σας, τη μητρική, να σας τα φέρουμε. Φέτος το φυλάδιο αυτό ακριβώς επικεντρώνεται στο θέμα της δεύτερης ευκαιρίας. Εντάξει περιλαμβάνει κάποια προφίλ από επιχειρηματίες που έχουν ε, ανακάμψει μετά από την πτώχευση και μοιράζονται μαζί μας τις ε, εμπειρίες τους. Είναι προφίλ διαφόρων ε, μεμονωμένων επιχειρηματιών που μπορεί να βρείτε μέσα σε αυτούς και κάποιον από την δική σας εκλογική περιφέρεια που έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία και μπορεί να σας πει και τα καλά και τα άσχημα της όλης διαδικασίας και τι ακριβώς χρειάστηκε να κάνουν για να επιβιώσουν και πώς κατάφεραν τελικά να επιμείνουν. Είναι πραγματικά κάτι που μας δίνει έτσι πολύ τροφή για σκέψη και μας εμπνέει. Ε, είναι δηλαδή πολύ προσωπικές ιστορίες και πολύ άμεσες αυτές οι ιστορίες μέσα στο φυλάδιο. Και αν θέλετε κι άλλα, ευχαρίστω να σας φέρουμε. So, ich darf mich herzlich bedanken. Jetzt noch Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Άλλη μία προσθήκη. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να προσθέσω κάποια σχόλια κι εγώ σε σχέση με τα όσα είπατε εισαγωγικά για την πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι περίπου 4 εκατομμύρια, μάλιστα 4,1 ε, θέσεις εργασίας δημιουργούνται από νέες επιχειρήσεις. Βεβαίω τα startups που θα τα βρούμε, ε, δεν τα πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Πρέπει να υπάρχουν νέοι επιχειρηματίε για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Χρειάζεται λοιπόν μια τέτοια ενισχυτική πολιτική και σε τοπικό και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό εδώ είναι ένα από τα στοιχεία. Σημαντικά, σημαντικό βέβαια, αλλά ένα. Υπάρχουν και άλλε πρωτοβουλίε που έχει πάρει η Κομισιόν, όπω α πούμε η προώθηση του προφίλ του επιχειρηματία γενικώ. Υπάρχουν ε, στη Δανία 80% του πληθυσμού που θεωρεί ότι οι επιχειρηματίες συμβάλλουν θετικά στον κοινωνικό ιστό. Στην Ουγγαρία το ποσοστό αυτό είναι μόλις 26%. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά και αυτό βεβαίω έχει συνέπειε και στην ετοιμότητα των νέων και στη διάθεσή του να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Δεύτερον, εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό σύστημα πολύ συχνά απομακρύνει τους πολίτες από οποιασδήποτε επιχειρηματικέ φιλοδοξίες, αντί να τους δίνει μια σωστή δίκαιη ευκαιρία για να καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει η επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες από την Κομισιόν για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητα στην, ε, και στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Έχουμε μια υψηλή ομάδα, ομάδα υψηλού επίπεδου, έχουμε, εκθέσει, έχουμε υποβάλει πολλές εκθέσεις, ε, κυρίως προς τις αρχές των κρατών μελών, ε, για τα υπουργεία τους, το Υπουργείο Οικονομικών και εκπαίδευση για να ενισχύσουν και αυτά το δικό του σύστημα. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, μπορούμε να, να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την γενική βελτίωση του περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα, για τις νέες επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άλλες εκθέσεις ε, που έχουν να κάνουν με τη μεθοδολογία που έχει ε, η Κομισιόν, με καλές πρακτικές, με συστάσεις, με στατιστικά στοιχεία, με την παρακολούθηση μετά την έναρξη αυτών των πρωτοβολιών. Γίνονται λοιπόν πολλά από την Κομισιόν και η Κομισιόν παρακολουθεί και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη. Οπότε εμείς ευχαριστώ να συνεχίσουμε μαζί σας τη συζήτηση για τέτοια θέματα εφόσον αυτά σας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, σήμερα θέλαμε να, να δούμε και τα θέματα και φρεγγιότητα κυρίω. Βεβαίως εδώ μιλούμε όμω για ένα πεδίο πολύ πιο ευρύ και νομίζω ότι όντω υπάρχουν πολλέ πτυχέ ενδιαφέρουσε. Θα πρέπει όντω να δούμε αν η πολιτική μα αυτή που ε, κάνουμε για τον πολίτη, βοηθάει τελικά τη ζωή του πολίτη ή μήπως του δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο. Καμιά φορά δεν είμαστε τόσο επιτυχείς. Εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Ποδηματάρχη το δυσκολευουμε ακομη περισσοτερο καμια φορα δεν ειμαστε τοσο επιτυχει εν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τους ε, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση που τουλάχιστον σε μένα επιβεβαίωσε αυτό που είπατε ότι αν ξέραμε τι ξέρουμε θα ξέραμε πολύ περισσότερα. Ε, θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση και να καταλήξω σε μια ερώτηση. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε για την ε, κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα, τις ε, διαδικασίες πτώχευσης μιας επιχείρησης, τις νοτροπίες κυρίως που υπάρχουν πίσω από αυτές τις διαδικασίες, το στίγμα, ε, το στίγμα το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δεν κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα στη δόλια πτώχευση και στην πτώχευση ε, που προκύπτει για λόγους ανεξάρτητους με τη θέληση του επιχειρηματία ε, το γεγονός ότι το στίγμα πηγαίνει στον επιχειρηματία και του στερεί τη δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας και όχι στην επιχείρηση που για χύψη λόγους δεν τα πάει καλά και όλα αυτά ε, για να το συνδέσω με αυτό αν ξέραμε τι ξέρουμε νομίζω ότι αναδεικνύουν την ανάγκη μιας συνέργειας δράσεων δηλαδή σε πολλαπλά επίπεδα ε, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα συνολικά ξεκινώντας από την πρόληψη όπως πολύ σωστά είπατε ε, και ε, φτάνοντας μέχρι την ριζική αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων και των αδυναμιών που περιγράψατε με πολύ γραφειρό τρόπο. θέλω να επισημάνω το εξής ε, ιδιαίτερα σήμερα σε συνθήκες μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην ευρωπαϊκή ένωση και στην ευρωζώνη ε, η ανάγκη να είμαστε πολύ ταχείς και πολύ κέρυοι στις παρεμβάσεις μας σε αυτό το τομέα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας εν γένει ένα τμήμα αυτής της ενίσχυσης ε, είναι η βελτίωση των διαδικασιών και των συνθήκων σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κήρυξη πτώχευση, καταπολέμηση του στίγματο, η ενίσχυση μέτρων δεύτερη ευκαιρία. Όλα αυτά είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα διότι ε, μόνο μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας θα βοηθήσουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και άρα την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, αυτό που παρατηρούμε όμως είναι ότι ειδικά στις χώρες της ευρωζώνης και της ευρωπαϊκής ένωσης που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες σήμερα εκεί ακριβώς τα προβλήματα της υποχώρησης της επιχειρηματικότητας και της κήρυξης διαδικασιών πτώχευσης πολύ συχνά ανεξαρτήτως της θέλησης και της βούλησης των επιχειρηματιών είναι ολοένα και πιο συχνά. Ε, άρα για να καταλήξω στο ερώτημά μου θεωρώ ότι όπως ακριβώς ε, λέμε για την οικονομική κρίση αυτή καθεαυτή όπως λέγαμε πριν από τρία χρόνια για τις τράπεζες υπάρχει ανάγκη δράσεων σε δύο επίπεδα θεσμικές δράσεις που αντιμετωπίζουν με ένα πιο μόνιμο τρόπο το πρόβλημα αλλά και δράσεις άμεσες έκτακτης ανάγκης που λέμε ε, που θα μπορούμε να τις υλοποιήσουμε αμέσως για να ανασχέσουμε όλες αυτές τις ε, ε, αρνητικές εξελίξεις που βαίνουν συνεχώς επιδεινούμενες σε σχέση με την επιχειρηματικότητα συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα περισσότερο στις χώρες που κατεξοχήν την έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Η συνάδελφο Χέρτσοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ του τρει ομιλητέ, τη Στέφανη, τον ε, κύριο Ρέστη και τον ε, πρόσωπο τη Κομισιόν. όντω, ε, έχουμε πολύ καιρό που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Εγώ Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη που επέλεξα να είμαι συγγήτρια για αυτό το φάκελο για τις μικρές επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά εξαιρετικό που βλέπουμε πώς από την ε, πρώτη στην ε, δεύτερη φάση έχουμε πολύ περισσότερες ε, επιχειρήσεις που ξεκινούν. Τώρα, για την πτώχευση, πολλοί μίλησαν για στίγμα, για στιγματισμό. Πρέπει να πω ότι πρόσφατα έμαθα τι σημαίνει στίγμα. Και επειδή είσαστε εδώ και οι τρει ε, έχετε συμμετάσχει στην ε, Σύνοδο Κορυφή πριν από ένα μήνα για τι μικρέ επιχειρήσει, ε, είχα την τιμή να είμαι και εγώ προσκεκλημένη από τον πρέσβη για τι επιχειρήσει από την Ουγγαρία για να μιλήσω για την πράξη για τι μικρέ επιχειρήσει. Πραγματικά δηλαδή πολύ σημαντική μέρα σήμερα για μένα και ο, πήρε ένα τηλεφώνημα από, από, έναν, από έναν άνθρωπο ο οποίος μου είπε ότι θα χάσει τη δουλειά του, ε, θα απολυθεί. Και είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ σήμερα τελικά να μιλήσω ακριβώς για αυτό το θέμα. Ήταν πραγματικά λοιπόν προσωπική εμπειρία μου όταν κατάλαβα τι σημαίνει στίγμα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η στιγμή είναι ιστορική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, τώρα, να γυρίσω στο θέμα. Είναι πραγματικά ζωτική σημασία να, μάθουν, να μάθουν οι πολίτες τι σημαίνει, ποιο είναι το, το, ποια είναι η απώλεια των επιχειρηματιών όταν πτωχεύουν και έχουν μετά δυσκολία να ξαναξεκινήσουν μια επιχείρηση. Αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν από μια εκπαίδευση. Όλες οι, ε, ε, όλα τους τα χρήματα τα έδωσαν σε μια, για να εκπαιδευτούν, επένδυσαν στην εκπαίδευσή τους και έχασαν και αυτό όσο δηλαδή ασχολούνται με την διαδικασία της πτώχευσης και δεν μπορούν να ξαναέρθουν στην ενεργοοικονομία και να αποδώσουν. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η γνώση που χάνεται. Και να θέσω ένα ερώτημα. Είπατε ότι από τέσσερα χρόνια θα γίνει τρία. Τα τρία χρόνια όμως είναι επίσης μεγάλη απώλεια. Κάνατε κάποια έρευνα για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα αυτά τα τρία χρόνια που δεν μπορούν να ξεκινήσουν μια δεύτερη δουλειά. Μπορούν να απασχοληθούν κάπου, μένουν άνεργοι, ε, με κάποιο τρόπο κάνουν, δουλεύουν στην μαύρη οικονομία, στην στη μαύρη αγορά. Τι ακριβώς κάνουν συγκεκριμένα, γιατί μιλούμε για ανθρώπους. Εγώ ως ε, σοσιαλίστρια πρέπει να πω ότι πολλές φορές ε, οι πολίτες εκπλήσονται όταν ε, μιλώ υπέρ των επιχειρήσεων. Αλλά είτε είναι μικρές επιχειρήσεις είτε είναι μεγάλες, δεν υπάρχει απασχόληση χωρίς αυτές. Οπότε πρέπει να δούμε και το θέμα της απασχόλησης, της πολιτικής απασχόλησης της Ευρώπης. Το άλλο θέμα που ήθελα να θίξω είναι ότι υπάρχει ένα ειδικό, ένας ειδικός τομέας όταν μιλούμε για την έναρξη των επιχειρήσεων στον τομέα της κοινοτομίας και της έρευνας γιατί η έρευνα δίνει μια τελ όταν ας πούμε υπάρχει έρευνα για ένα πολύ καταστροφικό προϊόν που θα μπει στην αγορά, ε, προφανώς επηρεάζει τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για αυτό, γιατί για μας την Επιτροπή Ήτρε, όταν παλεύουμε για να υπάρξουν κονδύλια για την έρευνα, για την κοινοτομία και προσπαθούμε να πείσουμε τους υπουργούς οικονομικών ότι αυτό δεν είναι κάτι χαμένο, είναι επένδυση στο μέλλον. Υπάρχουν πολλές ομάδες συμφερόντων που έχουν να κάνουν με την ε, εισαγωγή νέων και ε, καταξιωμένων ανθρώπων στην ε, αγορά εργασίας. Νομίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα μπορούσε να συνδέσει όλα αυτά τα δεδομένα και να εκπονήσει κάποιες πολιτικές. Αλλά αν αυτές οι πολιτικές είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό, τότε νομίζω ότι απλώς χάνετε το χρόνο σας. Προτείνω λοιπόν η Κομισιόν ίσως μα αποκοινούμε τους ευρωβουλευτές, να βάλει κάποια άρθρα για αυτό το πολύ συγκεκριμένο θέμα που μιλήσατε σήμερα σε μεγάλες εφημερίδες της Ευρώπης, έτσι ώστε οι α, α, επιχειρηματίες αλλά και οι πολίτες να μπορούν να τα καταλάβουν και ειδικά σε ένα τέτοιο περιβάλλον κρίσης. Όλοι σήμερα προσπαθούν να μειώσουν τις απώλειές τους. Και βεβαίω πάντα οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι αυτέ που υποφέρουν περισσότερο. Δε, τελευταίο μου σχόλιο. Όταν, προσπαθήσει, όταν προσπαθήσετε να, κάποιον να μάθει α, ποδήλατο, είναι πιο εύκολο να, να πείσετε κάποιον που έχει δοκιμάσει α, ή κάποιον που ε, δεν δοκίμασε ποτέ. Κάποιον δηλαδή που προσπάθησε να μάθει και απέτυχε ή κάποιον που δεν δοκίμασε ποτέ να μάθει ποδήλατο. Ευχαριστώ. Ο Πάολο Ρούμπιχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε είναι όταν ιδρύονται οι επιχειρήσεις, τότε γίνεται, χρειάζεται και ίδιο κεφάλαιο. Αν δηλαδή ιδρύει κάποιος μια επιχείρηση, θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει το απαραίτητο ίδιο κεφάλαιο. Ε, πολλές φορές ε, εδώ δίνονται ας πούμε κάποια δάνεια για να διευκολυνθεί η ίδρυση της επιχείρησης ε, και ουσιαστικά μετά το θέμα είναι να υπάρξει κέρδος. Η επιτυχία της επιχείρησης προκύπτει όταν κάποιος έχει υπηρεσίες ή πουλά υπηρεσίες ή προϊόντα οι οποίες όντως αγοράζονται και τα οποία όντως αγοράζονται από τους καταναλωτές. Γι' αυτό είναι σημαντικό να σκεφτούμε ε, το κέρδος που θέλουμε να επιτύχουμε. Να υπάρχουν δηλαδή περισσότερα έσοδα από ότι έξοδα έτσι ώστε να μην χρειαστεί να χάσει αυτό ο άνθρωπο την επιχείρησή του, να μην φορολογηθεί ε, άσκοπα, γιατί πραγματικά το κέρδος είναι η βάση του, της δημιουργίας του ίδιου κεφαλαίου και μετά να μπορεί κανείς να πάρει ένα δάνειο για να μπορεί να κάνει περαιτέρω επενδύσεις. Η, η φορολόγηση λοιπόν αυτών των κερδών είναι το ένα βασικό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε. Γιατί δεν υπάρχει μεγάλη δεν ρευστοποίηση στις επιχειρήσεις. Επίση, για τις απαλλαγέ. Αν, αν συγκρίνουμε λίγο τα πράγματα με την ε, Αμερική, για τέτοια μικρά ποσά στην Ευρώπη ε, μιλούμε για 300 ε, με 900 ευρώ. Στην, στη ΣΥΠΑ το ποσό αυτό είναι 5.000 5.000 ευρώ. Οπότε εκεί δεν μπορεί να υπάρξει φορολόγηση. Αν ας πούμε κάποιος ε, αγοράσει ένα αγαθό και μετά από κάποια χρόνια πρέπει να, το, πρέπει να απαλλαγεί γι' αυτό, ας πούμε όπως στην Αυστρία, όπου υπάρχει ε, χρονός παραγραφής 33 χρόνια, στη Γερμανία υπάρχει 50 χρόνια προθεσμία για, την, για αυτήν την απαλλαγή. Δηλαδή μια μια ε, επιχείρηση πρέπει να ε, προεπενδύσει για, για τα επόμενα 50 χρόνια και εντωμεταξύ σε αυτά τα 50 χρόνια φορολογείται ήδη το κεφαλαίο, το ε, κέρδος της. Πρέπει λοιπόν να δούμε πολύ συγκεκριμένα πώς θα καταφέρουμε οι επιχειρήσεις και ακριβώς τώρα σε καιρό κρίσης που δεν έχουν ίδιο κεφάλαιο να, να απαλλάσσονται από αυτή τη διαδικασία μπορούν, μπορεί να βρεθούν σε μια περίπτωση κρίσης, ε, ε, μέσω πρόθεσμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα περιβάλλον ευέλικτο για τις επιχειρήσεις. Αν απομακρυνθούν από τις ε, επιχειρήσεις, ουσιαστικά το κράτος είναι αυτός, αυτό που πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Και μετά καταλήγουμε σε, καταστροφές, σε καταστροφικές συνέπειες ό,τι αφορά το χρέος. Αυτό βεβαίως έχει επιπτώσει μετά και στην ε, οικονομία. Αυτή λοιπόν η άτεκτη στάση ε, δεν βοηθάει ούτε το ίδιο κεφάλαιο των επιχειρηματιών, ούτε, τις, ε, ούτε τους εργαζόμενους και επιβαρύνουν βεβαίως και το κρατικό χρέος και την ανεργία. Οπότε πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε καιρούς εργασίας για την δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να το σκεφτούμε. Σε τέτοιε μεγάλες, σε μεγάλες περιόδους επιτυχία και οικονομικής προκοπής ε, πρέπει να, επειδή ακριβώ υπάρχει μεγάλη οικονομική επιτυχία, να γίνεται μεγαλύτερη προσπάθεια σε ό,τι αφορά και τη φορολογία κτλ. Ενώ σε περιόδους ε, ύφεση και οικονομικής δυσπραγίας να είμαστε πιο ευέλικτοι και να μπορεί ο κάθε επιχειρηματία να παραμείνει στην επιχείρησή του. Επίση, για θέματα χρηματοδότηση. πρέπει να δούμε και τα χρήματα χρηματοδότηση και τα χρήματα φορολογία. Αν δεν τα λύσουμε αυτά τα θέματα γρήγορα, άμεσα, τότε η πίεση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και θα αρχίσουμε να μιλάμε για κατώτερους μισθούς και στο τέλος θα ε, εξαφαλιστεί και αυτή η ελάχιστη κοινωνική ασφάλεια που μπορούμε να δώσουμε στου πολίτε μα πρέπει να, είμαστε, να είναι συγκεκριμένος ο στόχος που έχουμε. Να έχουμε δηλαδή ο στόχο τους νέους που θέλουν να αναλάβουν την ε, ευθύνη μιας επιχείρησης, που θέλουν να ανοίξουν μια επιχείρηση και, που θέλουν να, και για κράτη που θέλουν να αναλάβουν την υποχρέωση των, της απασχόλησης των πολιτών τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα κίνητρα που δίνουμε στους νέους για να αναλάβουν ακριβώς την ε, ευθύνη μιας επιχείρησης. Ακόμη και αν αυτή η ε, επιχείρηση είναι μια ε, οικογενειακή επιχείρηση. Αν μπορεί να είναι ευέλικτη αυτή η οικογενειακή επιχείρηση και δεν μπορεί να χτυπάει σαν αντίχο γραφειοκρατία συνέχεια, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Χρειάζεται λοιπόν ε, μείωση της, της γραφειοκρατίας. Συγκεκριμένα συγκεκριμένες πολιτικές για την, και, για τους, και για τους μισθούς πρέπει να γίνει εξορθολογισμό, ε, δραματικός εξορθολογισμός αυτή τη στιγμή, γιατί ούτω ή άλλως σκοτώνουμε την, με αυτέ τι πολιτικέ και την ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Κέλλη έχει ζητήσει το λόγο. Ένα λεπτό θα σας δώσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο για απαντήσεις. Ένα λεπτό μονάχα. Αρκεί, αρκεί ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Πολ σε όσα είπε ε, σε όλα τα θέματα της πτώχευσης, της χρεοκοπίας ε, πρέπει να αλλάξει πλήρως η αντιμετώπιση μας και η προσέγγιση μας και δεύτερον να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την επιτυχία και την αποτυχία. Η, η αποτυχία στις ΗΠΑ αντιμετωπίζεται σαν μια μελλοντική επιτυχία. Οι αποτυχημένοι εδώ φέρνουν ένα στίγμα σαν να είναι παρίες και αυτό είναι ανθυγιεινό πιστεύω σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Θα έχουμε και επιτυχίες και αποτυχίες και τα δύο πρέπει να γίνονται αποδεκτά. Και προφανώς η εμπειρία των επιχειρηματιών είναι μάλλον η εμπειρία αποκτάται και μέσα από τις αποτυχίες και αν κάποιος ε, προσπαθήσει να κάνει κάτι την πρώτη φορά και αποτύχει τα διδάγματα αυτά θα τα ε, λάβει υπόψη του για τη δεύτερη προσπαθιά του άρα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο Λοιπόν, πέντε λεπτά η Κομισιόν, δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ, πέντε λεπτά. We will try to share. Θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που έθιξε η κυρία Χέρτσοκ για τον κίνδυνο. Πολλοί άνθρωποι όταν μιλάνε για την επιχειρηματικότητα λένε ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του επιχειρηματία είναι η ανάληψη κινδύνου. Και αυτό ε, είναι πολύ λάθος αντιμετώπιση. Είναι σαν να κάνεις bungee jumping χωρίς να είσαι δεμένος. Ε, το πρόβλημα είναι να έχουμε ένα κίνδυνο ο οποίος να είναι αποδεκτός. Και αυτό ισχύει και για την καινοτομία και για τις επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Ο κίνδυνος πρέπει να είναι διαχειρίσιμος. Γι' αυτό υπάρχουν έξι βήματα. Γιατί πρέπει να επενδύσεις περισσότερα χρήματα για να, γίνεις καλύτερη, για να κάνεις καλύτερη εκτίμηση και αξιολόγηση αξιολόγηση, θα πρέπει να δοκιμάσεις και να δεις και οι πελάτες σου τι λένε. Λοιπόν, πρέπει να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο. Και το καλύτερο βέβαια είναι να αποφεύγουμε τον κίνδυνο και όχι να τον αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο. Και η δεύτερη παρατήρηση όσον αφορά τον οικονομικό κίνδυνο αποτυχίας, όταν δείτε τα ατυχήματα τα αυτοκινητιστά, των αυτοκινήτων, οδικά ατυχήματα, ε, οι περισσότεροι λένε εντάξει δεν πειράζει, έγινε ατύχημα, η ασφάλεια θα πληρώσει. Πολλέ φορέ η ασφάλεια όμω πληρώνει πάρα πολλά χρήματα και στο κάτω-κάτω μπορεί να αγοράσει κανεί και καινούργιο αυτοκίνητο. Εδώ έχουμε σημαντικέ οικονομικέ συνέπειε. Όταν κάποιο επιχειρηματία ε, ε, όμω αποτύχει, ε, δεν, δεν γίνεται τίποτα και ίσως εκεί και τα, τα λεφτά τα οποία διακυβεύονται να είναι και λιγότερο. κανεί δεν ε, λυπάται τον κακόμοιρο επιχειρηματία. Ε, εγώ πιστεύω ότι ο επιχειρηματία πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη κατανόηση, διότι αυτό δίνει δουλειά και, στην, ε, και στου ε, συμπολίτε μα και γιατί προωθεί και την οικονομία. Τώρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη γιατί μας ενθαρρύνουν στο έργο μας. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσω το παράδειγμα των επιχειρήσεων που φορολογούνται συνεχώς και με επιπλέον φορολογία κτλ. Και υπάρχουν ε, κάποιες, ε, ε, κάποια παραδείγματα που ακριβώς αυτό δείχνουν. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα προσυζήτηση. Αν τώρα εσείς έχετε χρόνο και θέλετε να μπαίνετε και να βγαίνετε μέσα στην αίθουσα, τουλάχιστον κάντε το χωρίς να ενοχλείτε. Λοιπόν, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ξέρω ότι έχετε και άλλα θέματα να συζητήσετε. Λοιπόν, όπως σας είπα, ε, η ροή των κεφαλαίων είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ε, ε, κάτι που ανέφερε η κυρία Χέρτζοκ για την τριετή περίοδο. Δεν έχουμε το χρόνο να μπούμε σε πολλέ λεπτομέρειε, αλλά υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Το ένα είναι ο χρόνος για τις διαδικασίες πτώχευσης καθε, καθεαυτής και μετά τι γίνεται αφού εκαθαριστούν ε, τα χρέη. Ε, εάν μπορεί να ασκηθεί ε, δίωξη για να πληρώσει τα χρέη. Υπάρχει μια τριετής περίοδος και πιστεύουμε ότι όσο πιο σύντομη είναι η περίοδος τόσο καλύτερα. Δεν είδαμε από την πρακτική που παρακολουθήσαμε ότι το να αυξήσουμε την περίοδο δεν βοηθάει. Τώρα, για τις δικαστικές ε, ε, εξοδικαστικά μπορούν να ρυθμιστούν οι περισσότερε των περιπτώσεων. Δηλαδή, δεν μιλάμε για παραβίαση του ποινικού κώδικα ε, και νομίζω ότι εξοδικαστικά μπορεί να ρυθμίσουμε τις περισσότερες περιπτώσεις. Λοιπόν, σημειώσαμε τον επίγοντα χαρακτήρα του όλου θέματος και εδώ μιλάμε για ατομικές πτωχεύσεις, δεν μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις ή για τις τράπεζες, αλλά και εδώ είναι ένα παράδειγμα ε, όπου μπορούμε ε, να βρούμε μια γρήγορη λύση εξοδικαστικά. Κυρίες και κύριοι, λέει ο Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη. Εγώ γενικώ είμαι υπομονητικός άνθρωπος. Είμαι ήρεμος άνθρωπος. Αλλά πραγματικά είναι ντροπή, για να το πω απλά και ξεκάθαρα. Κάποιοι κύριοι και κάποιες κυρίες να μπαινοβγαίνουν μέσα στην αίθουσα και όλοι που είμαστε εδώ από τις 9 η ώρα το πρωί και ξεκινήσαμε τη συζήτηση, να μην μας αφήνετε να παρακολουθήσουμε. Δεν γίνεται. Μπορείτε να μπείτε με ησυχία να καθίσετε μέχρι να ξεκινήσουν οι ψηφοφορίε για να κουβεντιάσετε. Παρακαλώ, την κατανόησή σα για του υπόλοιπου συναδέλφου. Ξαναέχετε το λόγο, κυρία μου. I think we can conclude by saying that we Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενθάρρυνση. Χαιρόμαστε γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να, συζ... να προχωρήσουμε τη συζήτηση αυτή μαζί σας. Ε, μπορούμε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, ε, αλλά Νομίζω ότι θα πρέπει να το προωθήσουμε το θέμα γιατί είναι, έχει, είναι πήγον και χρειαζόμαστε τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πόρους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και τους βουλευτές. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εκπροσώπους της Κομισιόν κάναμε πραγματικά μια πολύ σημαντική συζήτηση ε, με πάρα πολλά στοιχεία. Ε, έχουμε ξεκινήσει από την ενεργειακή πολιτική, ε, ξεκινήσαμε σήμερα με τα οικονομικά θέματα, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον οικονομικό, οικονομικά ρευστό, ξεκινήσαμε να μιλούμε σήμερα το πρωί για την φερικιότητα των κρατών, για την πτώχευση και τι μπορούμε να κάνουμε. Πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο όλα τα στοιχεία είναι, ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η παρέμβασή σας. Σα ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας και βεβαίω σα υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε να το ε, συζητούμε. Ε, δεν είναι μόνο ένα το θέμα το σημαντικό που πρέπει να μας απασχολεί, είναι πολλά. Τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά ως πολιτικοί για να δώσουμε στις επιχειρήσεις μία ε, δυνατότητα να συνεχίσουν να υφίστανται, να μπορούν να λειτουργούν. Σα ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Thank you so much.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ζητώ συγγνώμη που έτσι εκνευρίστηκα λίγο, αλλά μερικές φορές είναι και κρίμα. Είναι κρίμα ως Επιτροπή να αναλαμβάνουμε, να καλούμε εδώ για να κάνουμε ακρόαση με κάποιους ε, εμπειρογνώμονες, με κάποιους ε, ε, εξπερ, ε, και όντω έχουμε τόσο πολύ λίγο χρόνο γιατί όλοι κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα να μην μπορούμε να τελικά να του ακούσουμε. Ε, ίσως λοιπόν θα πρέπει να δούμε αν πρέπει να ασχολούμαστε με λίγο λιγότερα πράγματα ε, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε όλα ταυτόχρονα. Ε, νομίζω ότι αυτό ήταν σημαντικό ε, και χάρηκα που τελικά καταφέραμε να το πράξουμε σήμερα, να έχουμε δηλαδή αυτούς τους εμπειρογνώμονες από την Κομισιόν εδώ. Κάποιος θέλει το λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ συνάδελφε. Συμμερίζομαι τα όσα είπατε κύριε Πρόεδρε, αλλά εγώ είμαι τακτικά παρόν εδώ στην Επιτροπή, αλλά σήμερα υπάρχει συμφόρηση γύρω από τις Βρυξέλλες και δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα στην πρωτεύουσα, γι' αυτό άργησα κατά μία ώρα. Ε, ήταν ένα θέμα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήθελα να λάβω το λόγο, δεν μπόρεσα να είμαι εδώ. Καταλαβαίνω τα όσα λέτε, αλλά ενοχλούμε πολύ περισσότερο από αυτοί που μπαίνουν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και εμποδίζουν τον εισηγητή να εκφραστεί με ησυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη στήριξη. Δεν ήταν προσωπικά τα σχόλια, εννοείται δεν είχα στόχο κανέναν, Απλώ ε, κάνει τόσο προσπάθεια η, Προεδρία, κάνει τόσο προσπάθεια το, η Γραμματεία να καλέσουμε του ε, εκπροσώπους και δεν του δίνουμε την απαραίτητη προσοχή. Ε, αυτό ένα με εκνευρίζει λίγο. Απλώ είπα, συνάδελφοι, αν μπορούμε, να το, αν μπορούμε να το βελτιώσουμε και αν τελικά θεωρείτε ότι μπορούμε, πώ θα το βελτιώσουμε. Λοιπόν, τελειώνει αυτό το σημείο, πάμε στι ψηφοφορίε. Έχουμε αρκετές ψηφοφορίες να διεκπαιρεώσουμε σήμερα και ξεκινούμε να διατηρήσουμε τη σειρά. Ο συνάδελφος Βιδέλκο άντρα είναι εδώ. Οπότε, να ξεκινήσουμε με τον χάρτη πορεία για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων αφρακούχων εκπομπών το 2050. Γνωμοδότηση. Έχετε, πρέπει να έχετε τα έγγραφα, πρέπει να έχετε τον κατάλογο της ψηφοφορίας. Ο κύριος ε, Πυρίλο είναι ο ε, εισηγητής. Να ξεκινήσουμε με την ε, ψηφοφορία. να βγάλω και εγώ την κάρτα μου. Ελπίζω να την έχετε όλη την κάρτα σας μαζί σας σήμερα, να την έχετε βάλει στο μηχανηματάκι. Λοιπόν, συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. 12 υπέρ, κατά, α, ε, συγγνώμη, από την αρχή. 12 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 σε δύο τμήματα. Α, μάλλον να το ελέγξουμε. Ωραία. Να το ελέγξουμε λοιπόν. Τη 12 ηλεκτρονικά. vote is open. Ένα λεπτό. Ε, πρέπει να, να ξεκινήσουν και τα μηχανήματα. Κοιμούνται μάλλον και αυτά ακόμα. Δεν δουλεύουνε. Κάτι ιδιαίτερο έχει αυτό το, αυτή η αίθουσα. Χθε είχαμε πάλι προβλήματα και το πρωί και το απόγευμα με, τα, με τους προτζέκτορες. Τώρα έχουμε πρόβλημα με τα μηχανηματάκια της ψηφοφορίας. Κάποιο φάντασμα κυκλοφορεί μέσα στην αίθουσα. Τι γίνεται, υπάρχει κάποιος τεχνικός εδώ να μας βοηθήσει. Yeah, yeah. But that needs more time. Παίρνει χρόνο το, το μηχάνημα. Λοιπόν, για να, να προσπαθήσουμε. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, ε, ας ξαναπροσπαθήσουμε. 12. Ποιος είναι υπέρ. 12 dafür. 1, Hatte hinein? Ja, die, also ist die Mehrheit dafür. Also, das ist, es ist etwas schwierig, meine Damen und Herren, wenn man aufzeichnet. Ναι, να, είναι λίγο δύσκολο όταν ανεβάζετε το χέρι σας, μετράμε, το κατεβάζετε και μετά το ξανανεβάζετε. Ε, καταλαβαίνετε, ή θα συμφωνείτε ή θα διαφωνείτε, δεν γίνεται ανάμεσα. Wer stimmt für den 12? Ποιος είναι υπέρ λοιπόν, Δο, τροπολογία 12.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 Ωραία. Απορρίφθηκε, απορρίφθηκε είχα, είχα δίκιο. Πάμε. Α, λειτουργεί τώρα. Όχι ακόμα. Μ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν μπορούμε να έχουμε σαφείς πλειοψηφίες. Λοιπόν, 13, πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 με προφορική τροπολογία και ψηφοφορία σε τρία όχι. Πρώτα η προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσει. Όχι. Ψηφίζουμε την ε, προφορική τροπολογία. Πρώτα. Ωραία. Πρώτα λοιπόν ψηφίζουμε την ε, προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Α, α, α τότε κατα... α, όλα καταπίπτουν. Εντάξει, τελειώσαμε. Όλα καταπίπτουν. Παρακάτω. 6. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 132, 123. Συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 60 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, απο, ε, εγκρίνεται. 34, όχι, πάει αυτή. 45 με προφορική τροπολογία υπέρ, όχι, όχι, τι θέλετε. Δεν υπάρχει προφορική τροπολογία. Είσαστε αντίθετοι με την προφορική τροπολογία. Α, μάλιστα. Ωραία, τώρα τι κάνουμε λοιπόν. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Ωραία. Οπότε ψηφίζουμε την 45 χωρίς την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την 45, τροπολογία 45 χωρίς την προφορική τροπολογία. Περιμένετε. Ο Βιντελ Κουάδρα έχει διαδικαστικό. Χωρί μικρόφωνο. Η ψηφοφορία της τροπολογίας 45 υπάρχει αντίρρηση από κάποιου από ό,τι κατάλαβα. Για αυτή την άκακη τροπολογία είναι δυνατόν για όνομα του Θεού. Γιατί να μην ψηφίσουμε την τροπολογία χωρίς την προφορική τροπολογία. εμεί δεν βλέπουμε το πρόβλημα, να ψηφίσουμε την τροπολογία με την προφορική τροπολογία. Είναι κρίμα. Γιατί συμφωνούμε όλοι. Ε, εντάξει, είναι λίγο άτεγκτη η στάση σας, συνάδελφε. Λοιπόν, ε, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Οι πράσινοι δεν συμφωνούν με την προφορική τροπολογία. Υπάρχουν κανόνε. Αυτοί δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε λοιπόν. Κρίμα. Οπότε ψηφίζουμε τη 45 χωρίς την ε, προφορική τροπολογία μπορεί να μην περάσει. Ψηφίζουμε τη 45 στην αρχική της εκδοχή. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αυτό ήταν. Να την ελέγξουμε, την, ε, την... Ε, ωραία, να ελέγξουμε μάλλον το μηχάνημα. Ψηφίστε αν είναι καλός ο καιρός. Ναι ή όχι. Ούτε ναι, ούτε όχι. Δεν ισχύει, δεν δουλεύει το μηχάνημα. Συνεχίζουμε με τη μέθοδό μας, χωρίς τεχνική. Θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει. Λοιπόν, 46. Υπέρ. Κατά. Α, ευχαριστώ. Ε, συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά. Ε, να, το, να το ξαναδούμε. 28 υπέρ. 28 υπέρ. Ψηλά τα χέρια σας. Κατά. Πρέπει να μετρήσουμε, λυπάμαι. Πρέπει να μετρήσουμε άλλη μια φορά. Πρέπει να ξαναμετρήσουμε. Δουλεύει? Δεν δουλεύει. Λοιπόν, ωραία, θα μετρήσουμε δύο λεπτά και τελειώνουμε. 28. Ποιο είναι υπέρ. Ψηλά τα χέρια τα κρατήστε τα μέχρι να μετρήσουμε. Gegenstimmen.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 15 ναι, 24 όχι. Κατα... Απορρίπτεται. 124 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέλος. Ψηφοφορία για το... για το σύνολο της ε, έκθεσης δεν έχουμε μηχανηματάκι, οπότε τα χέρια τα ψηλά, υπέρ, κατά, κατά, κατά. Ποιο είναι κατά. Κανεί δεν είναι κατά. Αποχέ. 5, 6. 6 απόχέ. 7 απόχέ. Οι υπόλοιποι υπέρ. Με μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη. Πάμε προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη. Μέχρι βέβαια να φτιαχτεί και το μηχάνημα, εμεί θα έχουμε τελειώσει με τι ψηφοφορίε. Ε, ε, συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. Η ε, συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, ε, ε, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 1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 κατά αποχές εγκρίνονται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τραν 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 12. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απο... Εγκρίνεται. NV8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές α, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 καταπίπτει. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται 102 υπέρ κατά Αποχέ, εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται 103 υπέρ κατά απόχέ, απορρίπτεται 106 καταπίπτει, 104 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά να το ελέγξουμε. 107. Έτοιμο το μηχάνημα. Ε, ορίστε, τα καταφέραμε. Συγχαρητήρια στους τεχνικούς. 107 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, το ΕΛΚ έχει έναν παραπάνω. Danke. Okay. 48 ψηφίσαντες 21 προς 26 απορρίπτεται. 108 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προσυμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ψηφοφορία για το σύνολο της πρότασης. Α, συγγνώμη, μου λείπουν κάτι σελίδες. Λοιπόν, NV1. Δεύτερο τμήμα μόνο ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στα, στις αιτιολογικές σκέψεις. Δύο. υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, citation 17. Συγγνώμη, συγγνώμη. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στα αισθητηλογικές σκέψεις. 2. Υπέρ. Το ίδιο, το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ. Είναι ο κατάλογος του ΕΛΚ. Ε, μάλλον κάποιες σελίδες λείπουν και από, και από άλλους, ε. Ναι, ούτε, ούτε εγώ ξέρω τι ψηφίζουμε, ναι. Και εμένα μου λείπουν οι σελίδες. Ναι, ναι, ναι. Ε, λυπάμαι, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε. Λείπει... Έχω την εντύπωση ότι τα, τα, στις ιδεολογικές σκέψεις είναι το θέμα. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε, πρέπει να ψηφίσουμε. Ναι, αλλά ε, τι να, πρέπει να ψηφίσουμε, δεν γίνεται. Ε, ε ναι, θέλουμε να τελειώσουμε, έτσι. Έχουμε πολύ λίγα, χωρί μικρόφωνο μιλάει η κυρία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε πολύ, ε, πολύ λίγε σελίδε. Για το 2 λοιπόν, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, ε, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχέ. Τι ήταν τώρα αυτό. Νομίζω απορρίπτεται. Νομίζω απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την, το σύνολο της ε, γνωμοδότησης. Interessante Methode. paar Seiten weniger. Als PPE eh zu viel. Ein, ja, jetzt eine Seite zu wenig, aber Έχουμε μια, μας λείπει μια σελίδα και έχουμε μια επιπλέον ψήφο από το ΕΛΚ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τέλος ψηφοφορίας. 48 ψηφίζοντες, 45 υπέρ, καμία κατά ψήφος και τρεις αποχές. Εξαιρετικά. Πάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Ευρώπη-Κίνα. Πάμε συμβαστική 1. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Ε, τροπολογία 7. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Α, να το ελέγξουμε. Μάλιστα. Να το ελέγξουμε. Παρακαλώ. 10. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το 10. Hey, the list is against. Ο, ο κατάλογος λέει κατά. Πάλι το ΕΛΚ έχει έναν παραπάνω. Εντάξει τώρα. Απορρίπτεται, εν πάση περιπτώσει. Συμβαστική 3, υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Ε, αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο... Σε ποιο νούμερο πάμε. Παράγραφος 3. Προφορική τροπολογία. Προφορική τροπολογία. Έχει κανείς αντίρρηση. Ωραία. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 σε δύο τμήματα. Να ελέγξουμε την 39, μάλιστα. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Είμαι καλός σήμερα. Ε, 40 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης άρχεται η ψηφοφορία Too much? No? It's okay. Vote Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Πάμε στην ε, έκθεση του κυρίου Μεζάρος. Πρώτη τελευταία ψηφοφορία. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 και 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά α, ξανά 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 να το ελέγξουμε μάλιστα να το ελέγξουμε την 4 παρακαλώ ψηφίζουμε την 4 Πέρας ψηφοφορίας και Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 και 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ. Κατά. Να το ξαναδούμε λίγο. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επτά. Με προφορική τροπολογία. Αντιρρήσεις. Όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Να το ξαναδώ. 49 υπέρ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 Αποχές. Απορρίπτεται. 23 υπέρ. Τι. Να ελέγξουμε. Μάλιστα. Να ελέγξουμε το... Το 21 καταπίπτει. 21 καταπίπτει. Το 22 θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. 22 λοιπόν. Να ελέγχουμε το 22. Board open. Closed and 21 to Απορρίπτεται 21 προς 28. 23 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Yeah, closed. Πέρας 49 ψηφίσατε, 45 προς 4. Ε, μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν, εγκρίνεται. Πάμε στο τελευταίο, δεν έχουμε άλλο ένα. Ε, ναι, πάμε στην έκθεση του Αλάζος Μεζάρος. Ξεκινάμε με την 1. Υπέρ, κατά, αποχές, α, απορρίπτεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6. Υπέρ, κατά,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 Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια σε όλους τους εισηγητές, τους κοιόδης, τους συνεργάτες και όλους τους υπόλοιπους που συμμετείχαν. Das war's. Wir machen weiter. Ωραία, συνεχίζουμε. Es gilt übrigens immer noch der Satz, bitte jetzt ruhig den Saal verlassen. Εξακολουθεί να ισχύει το διαλυθείτε ησύχος. My God, das was terrible, ne? Die Abstimmungsmaschine war echt ein Problem. Κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε. Πάμε στο περίφημο διάσημο σημείο, μια που είμαστε όλοι ε, εδώ στην αίθουσα, στο σημείο 14, ενωσιακό πλαίσιο εταιρική διακυβέρνησης, ε, συντάκτρια κυρία Λένα Κολάρσκα-Μπομπίνσκα. Πού είναι? Α, εδώ είναι. Η κυρία Μπομπίνσκα θέλει να μιλήσει, μπορείτε να την αφήσετε να μιλήσει. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Παρακαλώ, η κυρία Μπομπίνσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πράσινο, η πρόσινη βίβλο της Επιτροπής για την ε, διακυβέρνηση είναι ένα θεωρημένο πλαίσιο το οποίο πραγματικά για την ε, εταιρική διακυβέρνηση, το οποίο είναι ζωτική σημασία ε, για αυτή την ε, περίοδο την οποία ε, ζούμε. Πολλές επιχειρήσεις κατέρευσαν λόγω ακριβώς της λανθασμένης διακυβέρνησης. Η εταιρική διακυβέρνηση ανέκαθεν ήταν πάρα πολύ σημαντική, πόσο μάλλον τώρα. Το πλαίσιο το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή πρέπει να ενδυναμωθεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Συμπεριφοράς εφαρμόζεται και δεν θα πρέπει απλώς να παραμείνει γράμμα κενό. Θα πρέπει να υπάρξουν νέα μέτρα εφαρμογής ε, τα οποία θα λειτουργήσουν και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να σεβαστούν ε, τις διατάξεις του πιστεύουμε ότι ένας, ακούσα πολλούς που λένε ότι ο αυστριός έλεγχος είναι κατά της ελεύθερης εσωτερικής αγοράς. Δεν νομίζω όμως ότι ισχύει αυτό εδώ. Πολλές από τις προτάσεις μου ακριβώς θέλουν να ενδυναμώσουν τον έλεγχο και να γίνει πιο αυστηρή η εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο προτείνω έχει σαν στόχο να αυξήσει την ευθύνη των, των ε, διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων. Κάθε συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει τις κυρώσεις κτλ. Αλλά προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να πηγαίνουμε. Δεύτερον, προτείνω τα μέλη του Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου, να σέβονται κάποια κριτήρια γνώσεων ή να έχουν κάποια συγκεκριμένες, να, να αναλαμβάνουν κάποιους συγκεκριμένους δραστηριότητες. Προτείνω επίσης η Κομισιό να ε, εκδίδει ετησίως ε, μία έκθεση naming and shaming για τις περιπτώσεις μη εφαρμογής εταιρικής διακυβέρνησης. Ε, επίσης, προτείνω να να προωθούνται οι καλές πρακτικές, να ευαισθητοποιήσουμε τους ενδιαφερομένους για το πόσο σωστή και καλή είναι η διακυβέρνηση και κατά την άποψή μου θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, διότι πολλές φορές ε, πολλοί βρίσκονται σε πολλά διοικητικά συμβούλια Πολλές φορές έχουμε ένα άτομο το οποίο είναι παρόν σε πολλές εταιρείες. Αυτό θα πρέπει να περιοριστεί. Επίσης θα πρέπει να καταργηθεί η συμμετοχή των ανεπίσημων διευθυντών, των grey directors, που τοποθετούνται πολλές φορές από πολιτικά κόμματα ή από λόμπι. Επίσης, όλοι οι, θα πρέπει οι όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν κυρίως όσον αφορά την προστασία των, της μειοψηφίας. Και πρόσφατα η Κομισιόν, κυρία Ρέντινγκ, ζήτησε να υπάρξει ε, η, μια ελάχιστη γυναικεία παρουσία στα συμβούλια. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, είναι αμφιλεγόμενο. Εγώ συμφωνώ πάντως. Πιστεύω θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα δύο φύλλα όσον αφορά τον τρόπο τον οποίο εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο και αυτή ακριβώς η άποψή μου αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Μπομπίνσκα. Ο κύριος Ντεάντζελης έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σημερίζομαι και την δουλειά που έχει κάνει και την ε, προσπάθεια της ε, συναδέλφου. Είναι μια καλή πρόταση, πάρα πολύ ισορροπημένη, που ασχολείται με ένα πρόβλημα, με ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό, ε, κυρίως τώρα με την κρίση, οικονομική κρίση την οποία να περνάμε, η οικονομική κρίση η οποία πιέζει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το θέμα επομένως της διαχείρισης των κινδύνων είναι πολύ σημαντικό και η κακή ε, ε, διαχείριση των κινδύνων είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί λύση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε καλές πρακτικές, Χρειαζόμαστε μια καλή διακυβέρνηση, μια καλή εταιρική διακυβέρνηση. Η πρόταση της ε, κυρίας Μπομπίνσκα ε, περιλαμβάνει κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ απτά και συγκεκριμένα. Είμαι πεπισμένος ε, για την ε, σημασία του θέματος, γι' αυτό ε, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη για διαφάνεια, την αρχή της ευθύνης και την σύγκρουση συμφερόντων. Αυτά για μένα είναι τρία θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Κυρίως αναφορά την εμπιστοσύνη την εμπιστοσύνη και της αγοράς. Επίσης είναι σημαντικό το σημείο όπου αναφέρεται η ισότητα των δύο φύλων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με βρίσκει σύμφωνο. Πιστεύω επομένως ότι χρειάζονται νέα μέτρα, χρειάζονται νέα εργαλεία να επικαιροποιηθεί το όλο πλαίσιο, ε, έχουμε, να έχουμε κώδικα συμπεριφοράς, να έχουμε κυρώσεις, αλλά ταυτόχρονα να επιβραβεύουμε και αυτούς ε, που εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις της κυρίας Μπομπίνσκα. Ο συνάδελφος Βέμπερ έχει το λόγο. Oui, <clears throat> Ναι, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ε, έκθεση αυτή, έκθεση η οποία νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα επίκαιρη. Οι επιχειρήσεις ε, έχουν, την τάση εδώ και 15 χρόνια περίπου να προωθούν, να θέλετε, τους μετόχους εις βάρος άλλων εταίρων που είναι παραδείγματος χάρη οι εργαζόμενοι στα διοικητικά συμβούλια πιστεύω ότι η εκπροσώπηση των εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και όχι μόνο στα συμβούλια επίβλεψης. Ίσως επομένως το κείμενό σας θα έπρεπε να ενδυναμωθεί σε αυτό το σημείο κατά τα λοιπά. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών και ίσως εκεί θα έπρεπε το κείμενο να είναι πιο δεσμευτικό, διότι εάν δείτε ποιες είναι οι πρακτικές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα στην Νορβηγία, ε, θα δείτε ότι παντού όπου ε, επιβλήθηκε, ε, αν θέλετε, η παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Γιατί αν τα αφήσουμε όλα στην καλή θέληση, στην λογική και στον, και στον αυθόρμητο χαρακτήρα ας πούμε, των υπευθύνων, τα αποτελέσματα δεν θα είναι λαμπρά. Πρέπει να υπάρχει και ένα υποχρεωτικό χαρακτήρα, ένα δεσμευτικό χαρακτήρα για να γίνει κάτι. Όπω και στην πολιτική για να, σπάσει αυτό να σπάσουν τα εμπόδια. Και στην Νορβηγία είδαμε ότι και όσον αφορά την οικονομική συμπεριφορά και απόδοση των εταιριών, η, η παρουσία των γυναικών ε, ήταν θετική. Επομένως δεν είναι απλώς και μόνο ένα θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης ε, ή αστικής ευθύνης τέλος πάντων, είναι και ένας ε, στόχος αποτελ... Ε, οικονομικής αποτελεσματικότητας η παρουσία των γυναικών. Κύριος Χόκμακα, ευχαριστώ πρόεδρε και ενας στοχος αποτελ οικονομικης αποτελεσματικοτητας η παρουσια των γυναικων κυριε σχοτμακα ευχαριστω προεδρε και ευχαριστω και την εισηγήτρια για την έκθεσή της για ένα δύσκολο θέμα και είναι δύσκολο, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με διαφορετικές παραδόσεις, με διαφορετικές νομοθεσίες ε, στις διάφορες χώρες ε, και όλοι έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ε, στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι εταιρείε δέονται μεταξύ τους. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικό, ένα σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε, είναι ότι εάν δεν υπογραμμίσουμε την ευθύνη των ιδιοκτητών δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια νομοθεσία, στο μέλλον τουλάχιστον, που να υποσκάπτει την ε, ευθύνη των ιδιοκτητών, για δύο λόγους. Διότι αν θέλουμε να κάνουμε πιο εύκολο τον τρόπο που θα αναπτύσσονται οι εταιρείε, οι επιχειρήσει στην Ευρώπη, θα πρέπει να ε, συνειδητοποιήσουμε τις ευκαιρίες που έχουν οι ιδιοκτήτε. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε κιόλας και για την ευθύνη των εταιριών, τότε η ευθύνη θα πρέπει να στηρίζεται στις αποφάσεις των ιδιοκτητών. Και η άποψή μου είναι, διαβάζοντας εδώ τις και κοιτάζοντας τις διάφορες παραδόσεις που ισχύουν ε, στις ε, χώρες μας, ε, βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες οι ευθύνε των ιδιοκτητών είναι λίγο ασαφείς, όπου τα διοικητικά συμβούλια είναι κλειστά έστω και αν το ξέρουν όλοι ότι είναι ευθύνη των ιδιοκτητών να πούνε ναι ή όχι, η συζήτηση για το νέο συμβούλιο και η επιλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ε, με κλειστές τις πόρτες. Επομένως πιστεύω ότι το μήνυμά μας προς την Κομισιόν είναι ότι χρειαζόμαστε διαφάνεια δεν χρειάζεται να έχουμε ένα μοντέλο ενιαίο, διότι ούτως ή άλλως το εταιρικό δίκαιο διαφέρει από χώρα σε χώρα. Είναι ε, δύσκολο να πάρουμε όλα τα εταιρικά δίκαια και να μετά σε όλα αυτά τα εταιρικά δίκαια να επιβάλλουμε μια ενιαία εταιρική διακυβέρνηση, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις παραδόσεις και τον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργούν και δημιουργούνται οι επιχειρήσεις. Αν δείτε τι γίνεται σε δικιά μου τη χώρα. Μπορούμε να έχουμε μέλη σε ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο να έχουν διαφορετικές εμπειρίες. Και αν δούμε τις μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε άτομα τα οποία ε, είχαν εμπλακεί στην, ε, ενεργά στη διαχείριση κάποιων ε, εταιριών και μετά ήταν μέλη σε άλλα διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή και καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να είναι, αν πούμε, ας ότι πρέπει να είναι μόνο μέλη σε δύο διοικητικά συμβούλια, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να επωφεληθούμε από τον επαγγελματισμό και την εμπειρία που έχει κάποιο. Αλλά το πιο βασικό σημείο για μένα είναι ότι είναι ευθύνη των ιδιοκτητών και είναι δύσκολο να αποφασίσουμε από την ευρωπαϊκή σκοπιά τι θα γίνει σε διαφορετικές οικονομίες που έχουν διαφορετικές δομές. Επομένως πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε την διαφάνεια και την ευθύνη των ιδιοκτητών. Και εδώ όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων, πιστεύω ότι ζούμε μια αλλαγή και η εμπειρία που έχουμε εμείς είναι αντίθετη από, αυτούς τους, από αυτή των Νορβηγών. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε δύο διαφορετικές κατηγορίες στο Συμβούλιο, διότι με κάθε σεβασμό για τις προτάσεις ε, της Πράσινης Βίβλου, κατά την άποψή μου αυτό είναι παλιωμοδίτικο. Αυτό ίσχυε πριν από πολλά χρόνια, όταν βάζαμε σε διαφορετικές κατηγορίες άντρες και γυναίκες. Ε, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε αντίθετα την ευθύνη των εταιριών να λάβουν υπόψη τους όλα τα προσόντα που είναι διαθέσιμα. Ε, και εκεί λαμβάνουν υπόψη και οι γυναίκες και οι άντρες και αλλά όχι μόνο αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να έχουμε ε, ένα μοντέλο το οποίο να επιβληθεί στις διάφορες επιχειρήσεις, στις διάφορες χώρες, διότι εκεί το εταιρικό μοντέλο είναι διαφορετικό. Και υπογραμμίζω για άλλη μια φορά την ευθύνη των ιδιοκτητών, διότι δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να ε, αφαιρείται η τελική ευθύνη από τους, ε, από τους ιδιοκτήτες και οι ιδιοκτήτες να μην έχουν πλέον ευθύνες. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Χένεν. Κύριε Πρόεδρε, επανέρχομαι στην παρέμβαση του προλαλήσαντος ότι θα πρέπει να εμπλουτιστούμε από, την διαφορά, που, από τις διαφορές για να προτείνουμε νέες και πιο εμπλουτισμένες απαντήσεις στην κοινωνία. Έχουμε διαφορετικές εμπειρίες, ε, εμπειρίες μας όλοι μας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να αποφασίσουμε έναν κανόνα με τον οποίο να ταυτίζονται όλοι στην Ευρώπη. Γιατί αλλιώς ε, τι θα έχουμε, ε, ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή σε εθνικό επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο, σε παγκόσμιο επίπεδο όπου ε, ο καθένας ε, θα λειτουργεί με τον δικό του τρόπο. Έχουμε ομίλους ας πούμε στη Γαλλία που έχουν έρθει ε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν φρικτές συμπεριφορές απέναντι στους εργαζομένους, αλλά όχι μόνο και απέναντι σε όλη την κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι μια εταιρεία θα πρέπει να είναι υπόλογη απέναντι και στους εργαζομένους της και στην κοινωνία, γιατί χρησιμοποιεί την κοινωνία για να προχωρήσει. Επομένως, αυτές τις εταιρείες θα πρέπει να τους ζητήσουμε ε, να κάνουν μια ελάχιστη προσπάθεια ε, για να έχουν σωστές σχέσεις με την κοινωνία, τουλάχιστον ισότιμες ε, σχέσεις με την κοινωνία. Για τις γυναίκες τώρα ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και οι Εθνικές Νομοθεσίες έχουν προβλέψει οι εργαζόμενοι να είναι ενημερωμένοι, αλλά πολλές φορές ε, για να ενημερωθούν, είναι υποχρεωμένοι να, πάνε στην, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να αποκτήσουν τις ελάχιστες πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες για να προχωρήσουν. Δηλαδή ακόμα και αν η νομοθεσία το προβλέπει, πολλοί υπεύθυνοι εταιριών δεν περιμένουν να φτάσει η υπόθεση στα δικαστήρια για να δώσουν τα, τα χαρτιά, τα, οποία, τα έγγραφα τα οποία πετούνται. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι Πολλές φορές ε, ε, αυτό το θέμα των ε, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη τα οποία εμφανίζονται σε πολλά διοικητικά συμβούλια, αυτό είναι λίγο επικίνδυνο κατά την άποψή μου. Ε, γιατί δημιουργούνται διάφορες ε, πλειοψηφίες ε, για να μπλοκάρουν τις, τη λειτουργία κάποιων εταιριών. Λοιπόν, δεν πρέπει να μετουσιώνουμε, αν θέλετε, τον, τον νόμο. Στην πρώτη συζήτηση, στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας μιλήσαμε για την πτώχευση. Τώρα η πτώχευση και η χρεοκοπία χρησιμοποιείται από μεγάλες επιχειρήσεις, τελείως, κυρίως για τις υπεργολάβους, για να σπάνε τις τιμές. Ε, θα πρέπει να δούμε τι αυτό το οποίο επιτρέπει ο νόμος πώς χρησιμοποιείται για να καταλήξουμε σε ένα θέμιτο ανταγωνισμό. Γι' αυτό θα πρέπει ο νόμος να εφαρμόζεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ναι, ευχαριστώ. Να πω ότι διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί ε, ως πολιτικοί, να μην ε, γίνουμε έτσι εμείς που θα καλλιεργούμε την κουλτούρα της επιχείρησης γιατί η συνένεση που υπάρχει στην κοινωνία ε, και ελπίζω να υπάρχει και εδώ είναι το πώς διοικείται μια επιχείρηση είναι θέμα της επιχείρησης. Και εμείς απλώς πρέπει σε πολιτικό επίπεδο να, εξι, να, εξε, να αξιολογήσουμε ποιες είναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αναλαμβάνει μια επιχείρηση. Ως πολιτική λοιπόν ε, νομίζω ότι θα γίνουμε τελείως αναξιόπιστοι γιατί οι πολιτικοί ήταν και αυτοί που ξεκίνησαν, που δημιούργησαν την κρίση χρέους στην Ευρώπη και που φτάσανε τα πράγματα εδώ που φτάσανε. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, διστακτικοί. Ίσως ε, βεβαίως με να αλλάξει και το γενικό, έτσι, γενική ε, γεωγραφία των ε, επιχειρήσεων στην Ευρώπη με τον νέο αυτό καναόνα. Βεβαίως έχουμε και, τους, και τις ποσοστώσεις για, τις, για την ύπαρξη των δύο φύλων στις επιχειρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε και ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών. Τι λειτουργεί κάτι και πού λειτουργεί καλά και τι λειτουργεί κάτι και πού λειτουργεί άσχημα. στη Γερμανία σήμερα εμείς ε, έχουμε κάποια ε, ε, διοικητικά συμβούλια τα οποία βεβαίω έχουν μία ποσόστοση γυναικών αντρών και αντιστοίχω λαμβάνουν τι αποφάσει τους. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε αν η Ευρώπη θα αναλάβει όχι ένα, αυτό το παράδειγμα. Και να τονίσω επίσης ότι οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όταν είναι πολύ μεγάλες, δεν έχουν μόνο στόχο τις ανάγκες των μετόχων. Προφανώς, ε, με, εκεί κινούμαστε σε ένα πεδίο έντασης μεταξύ του σωστού πλαισίου πολιτικής, μεταξύ ε, γενικής αποδοχής, αυτού δηλαδή που θέλουν οι πολίτες και αυτού που θέλουν οι μέτοχοι. Οπότε η γενική αυτή θεώρηση ότι οι επιχειρήσεις, ακόμα και όταν είναι μεγάλες, μόνο και αποκλειστικά σκέφτονται το κέρδος ε, και, και μόνο αυτό, ε, νομίζω ότι μάλλον ε, ήταν ε, ε, θέμα παλαιότερων εποχών και δεν ταιριάζει τη σημερινή εποχή. Οι εταιρείε πάντα υπόκεινται σε πολύ αυστηρή κριτική από την κοινή γνώμη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μην, να μην δώσουμε έτσι, τέτοια δικαιώματα και εμείς εδώ να μην ε, υπερρυθμίσουμε λοιπόν τα πράγματα για κάποιον που θέλει να δημιουργήσει μια ε, εταιρεία. Δεν νομίζω ότι θα κάνει αυτό πολύ καλύτερη την Ευρώπη, απλώς θα την κάνει πιο γραφειοκρατική. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, η Κομισιόν θέλει κάποιος να απαντήσει. Υπάρχει κάποιος εδώ από την Κομισιόν. Θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Η Κομισιό μόλις δημοσίευσε πριν από μερικές μέρες ένα feedback statement μετά την φάση των διαβουλεύσεων. Νομίζω ότι η ποιότητα των προτάσεών σας θα είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να εξετάσουμε. Τα μέλη του Κοινοβουλίου εξάλλου το είπαν σήμερα το πρωί. Βρισκόμαστε σε ένα σύστημα με διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικές πρακτικές Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας. Πολλά από αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα λάβουμε υπόψη και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων για να παράγουμε ένα σύστημα που θα μπορεί να λειτουργήσει στο επίπεδο της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπομπίνσκα, μήπως θέλει το λόγο και πάλι, παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω που στην εισήγησή μας βρήκατε την δήλωση ότι οι εταιρείε προσανατολίζονται μόνο προς το κέρδος. Δεν είναι κάτι ε, που θέλησα να αποτυπώσω. Βεβαίω, απευθυνόταν σε συνάδελφο και όχι σε μένα αυτή η παρατήρηση. Πάντως δεν νομίζω ότι έτσι είναι η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι η οικονομία πρέπει να αφαιθεί μόνη της επειδή οι επιχειρήσει και οι ιδιοκτήτε τους μπορούν να ρυθμίσουν τα πάντα. Αυτό δεν ισχύει και το βλέπουμε σαφώς τώρα. Βλέπουμε ότι όλη η ομάδα των ε, επιχειρήσεων και των οικονομικών οργάνων υποφέρουν, βλέπουμε τον κατακαιρματισμό, λέτε ότι οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι. Ωστόσο, στον σύγχρονο καπιταλισμό το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης ή δύο ιδιοκτήτες. Δεν υπάρχει σαφές καθεστώς ιδιοκτησίας. Η ιδιοκτησία είναι πάρα πολύ συχνά κατακαιρματισμένη, υπάρχουν μερικοί συγκαλυμμένοι μέτοχοι, δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι νομίζω μια λέξη κλειδί, είναι αυτό που θέλουμε να έχουμε περισσότερο από όλα. Καμιά φορά οι ιδιοκτήτες χρειάζονται βοήθεια για να περιορίσουν ορισμένες πρακτικές που κατά τη γνώμη μας δεν είναι οι κατάλληλες. Δεν προσπαθούμε να τα κωδικοποιήσουμε όλα. Μιλάμε για ορισμένες κατευθύνσεις, για δράσεις, για μέτρα. Σχετικά με τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να μιλάμε πολύ για τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά αν δεν υπάρχουν ποσοστώσεις, δεν θα υπάρχει ισορροπία μεταξύ των φύλων και καμία επίπτωση στην πράξη. Βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές παραδόσεις, τις απαιτήσει της ελεύθερης αγοράς. Δεν πρέπει να επιβάλλουμε υπερβολική πειθαρχία. Ωστόσο, ορισμένα πράγματα Ορισμένες δράσεις ε, χρειάζονται υποστήριξη ή προτάσεις από πλευράς μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, να πω, 5η, ε, Όποιοι έχετε ακόμα να υποβάλλετε τροπολογίες, μέχρι την 5η 12 το μεσημέρι. Πάμε στην προστασία των υποδομών. Και επόμενος, επόμενο βήμα για την επιτεύγματα και επόμενα βήματα προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Εισηγητής ο κύριος Κάλφιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, με συγχωρήσετε, δεν έχω ετοιμάσει το έγγραφο συζήτησης. Θα πρότεινα στους κοιόδης εισηγητές ε, σχέδια ε, τις επόμενες μέρες για να συζητήσουμε το κείμενο για την εισήγηση. Θέλω να προτείνω διάφορα πράγματα που θα έπρεπε να περιληφθούν ε, σε αυτή την έκθεση. Ποια είναι η λογική. Η Επιτροπή έχει εκδώσει δύο ανακοινώσεις ε, σχετικά με την προστασία των κρισίμων υποδομών το 2009 και το 2011 και υπάρχει ένα σχέδιο για το πρόγραμμα δράσης CIP. Εκτός από αυτό, σε διάφορα ε, έγγραφα νομοθετικά και μη, η κυβερνοασφάλεια αναφέρεται σε διαφορετικά πλαίσια. Ε, ένας φόρος, ε, μια οδηγία για τον φόρο, για τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, η ψηφιακή ατζέντα, έκθεση πρωτοβουλίας. Έχουμε σε διαφορετικά έγγραφα διάφορες πληροφορίες και διάφορες διατυπώσεις τα οι οποίες αναφέρονται στην ασφάλεια, Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κατανοούμε ε, τις τεχνολογίες πληροφορίας ε, και με, ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Ό,τι και να κάνουμε η νομοθεσία θα υστερεί α, της τεχνολογίας, κάτι που είναι προφανές, δεν χρειάζεται να αναπτύξω το θέμα. Και το δεύτερο είναι ότι ο κλάδος θα περιμένει τις αντιδράσεις των θεσμικών οργάνων. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας και να δεχθούμε ότι οι τεχνολογίες αναπτύσσονται ταχύτατα και ο κλάδος ο ίδιος ασχολείται με την ασφάλεια στον κύβερνο χώρο. Τα όργανα θα πρέπει ίσως να εναρμονίσουν τις διαδικασίες και να λάβουν προληπτικά μέτρα. Υπάρχουν δύο ε, προκλήσεις σχετικά με τον χώρο και το διαδίκτυο. Τα εγκλήματα στον χώρο που είναι κοινά, η πορνογραφία, ε, η υποκλοπή, το hacking ε, των τραπεζικών λογαριασμών, παραβίαση των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η νομοθεσία ισχύουσα πρέπει να εφαρμόζεται στο διαδίκτυο και έχουμε ήδη πολύ καλά παραδείγματα καλής συνεργασίας στην Europol για την δίωξη τέτοιων αδικημάτων. Απλώς πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ισχύουσα νομοθεσία καμιά φορά εφαρμόζεται σε διαφορετικό χώρο που είναι ε, το διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος. Έχουμε και νέες προκλήσεις που ε, εμφανίζονται σε σχέση μόνο με το περιβάλλον ε, του κυβερνοχώρου. Έχουμε τα botnets, αυτά τα δίκτυα ρομπότ, τα οποία βρούν και αυτές είναι απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που είναι στενά συνδεδεμένες με το περιβάλλον του διαδικτύου. Εδώ δεν έχουμε ε, τρέχουσα νομοθεσία και θα πρέπει να σκεφτούμε τουλάχιστον κάποιο πλαίσιο για να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα. Ένα καλό παράδειγμα είναι η πρόταση της Επιτροπής για τις επιθέσεις στις ε, πληροφορίες. Ποινικοποιούνται τα botnets, τα ρομπότ αυτά και ε, θα πρέπει να συγκλίνουν ε, οι νομοθεσίες των διαφόρων κρατών μελών. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια συνεκτική προσέγγιση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Όταν αναφερόμαστε σε συνεκτική προσέγγιση, νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική που να θέτει το γενικό πλαίσιο για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δρά στον τομέα της ασφάλειας και να λάβουμε υπόψη νέες εξελίξεις, τη χρήση cloud, computing, ε, δικτύων, εφιών δικτύων κλπ. Ταυτόχρονα η στρατηγική αυτή θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ανθεκτικό σύστημα στον κυβερνοχώρο. Δεν είναι τόσο για την προστασία εναντίον μεμονωμένων επιθέσεων, αλλά ε, για να βεβαιωθούμε ότι ε, είναι βιώσιμα τα συστήματα ε, και ανθεκτικά επειδή είναι θέμα ορισμών επίσης που τίθεται όταν ε, μιλάμε για την προστασία κρισίμων ε, σημαντικών υποδομών, δεν έχει ακόμα δοθεί ορισμός τι είναι κρίσιμη δομή υποδομή, αν συμφωνούμε για τα ηλεκτρικά δίκτυα, για τα δίκτυα ε, ίδρευσης. Δεν συμφωνούμε για την υποδομή πληροφοριών και θα πρέπει να εμβαθύνουμε στο διάλογο με τους εμπλεκόμενους, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον ίδιο τον κλάδο για να δημιουργήσουμε ε, κανονισμούς ε, για τον χώρο αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει ανοιχτή προσέγγιση όταν το πλαίσιο αναπτυχθεί, να έχουμε διαβουλεύσεις ε, με τους ενδιαφερόμενους. Η Κομισιό άρχισε μια καλή άσκηση για να αναπτύξει την στρατηγική του cloud computing ε, για να διαβουλευθεί με τα εμπλεκόμενα μέρη. Θα πρέπει αυτό να διευρυνθεί όταν ε, θέλουμε να θέσουμε ένα γενικό πλαίσιο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Θα υπάρξουν προσπάθειες για να τεθούν ελάχιστα πρότυπα ε, περιβαλλαμβάνοντας ε, τις βέλτιστες πρακτικές, την διαλειτουργικότητα και ίσα η υπηρεσία ασφαλείας είναι ενεργός εταίρος και έχουμε μια έκθεση η οποία εξετάζεται στην Επιτροπή μας σχετικά με την εντολή της ΦΙΣΑ και θα πρέπει να περιληφθεί σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης δύο ή τρία σημαντικά πράγματα όταν αναπτύσσουμε το γενικό πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα με ε, τις ευαίσθητες πληροφορίες αν υπάρχει αντίθεση από κράτη-μέλη να προχωρήσουν με τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον ε, κυβερνοχώρο. Αυτό έχει να κάνει με την ε, χρήση ευαισθήτων πληροφοριών για διάφορες χώρες. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να ανανεωθεί τώρα, διότι δεν είναι μόνο η πρόσβαση στις ευαίσθητες πληροφορίες, αλλά πρόκειται για την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για ανθεκτικές υποδομές. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσελκύσει πολύ καλύτερα την προσοχή των κρατών μελών. Το δεύτερο θέμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν θα προετοιμάσουμε το γενικό πλαίσιο είναι η ελευθερία ανάπτυξης τεχνολογιών. Πολύ συχνά εδώ προσπαθήσαμε να περιορίσουμε ε, την χρήση τεχνολογιών και διαδικτύου, διότι δεν ξέρουμε πώς να προλάβουμε την κακή χρήση αυτών των ε, τεχνολογιών. Θα πρέπει μάλλον εδώ να υιοθετήσουμε μια στρατηγική και πολιτική που να επιτρέπει ακόμα και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τεχνολογιών και τη χρήση τους ε, για να έχουμε ασφαλή κυβερνοχώρο. Και τέλος θα πρέπει να έχουμε προσβασιμότητα ε, και εύκολη δυνατότητα. Αυτές τις αρχές θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη όταν αναπτυχθεί η στρατηγική. Και πάλι σε σχέση με το γενικό πλαίσιο μπορεί να υπάρξουν πολλά θέματα σε σχέση με την παιδεία, την κατάρτιση, ε, του πλωτισμού και όσων ασχολούνται με τον κυβερνοχώρο. Το δεύτερο πράγμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει, εκτός από το γενικό πλαίσιο, είναι ο μηχανισμός εφαρμογής των πολιτικών. Έχουμε ήδη την ε, υπηρεσία αυτή για την οποία μίλησα. Έχουμε την συνεργασία με την Europol, αλλά θα πρέπει ακόμη να δημιουργήσουμε πιο ισχυρούς μηχανισμούς για να εφαρμόσουμε τους, ε, τα γενικά μέσα, τα ευρύτερα μέσα για την ε, κυβερνοασφάλεια και να συζητήσουμε ευαίσθητα θέματα, παραδείγματο χάρη αν θα υπάρχει υποχρέωση ε, δημόσιας κοινοποίησης των κυβερνοεπιθέσεων. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που συνδέεται επίσης με το μηχανισμό εφαρμογής. Και τέλος, αυτό που θα πρότεινα να έχουμε σε αυτή την έκθεση είναι το θέμα που σχετίζεται με την διεθνή συνεργασία και αντιπροσώπευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, εφόσον η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο συνδέεται με τη διεθνή συνεργασία. Έχουμε μερικά θετικά βήματα από, ε, από πέρσι όταν περιελήφθηκε η ασφάλεια αυτή στον διατλαντικό διάλογο και δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένε Πολιτείε για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αλλά θα πρέπει να διευρύνουμε τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαδραστική ε, δραστηριότητα με άλλες χώρες για να έχουμε ισχυρότερη διεθνή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω με μερικά διαδικαστικά θέματα για να προτείνουμε στις πολιτικές ομάδες τους σκιώδεις εισηγητές ένα κείμενο που θα μπορούμε να συζητήσουμε και ίσως θα μπορούσαμε ίσως να, να θεωρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και να έχουμε του χρόνου, ίσως τον Ιανουάριο, την, το κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Φανίστελ Ροϊ, ο επόμενος. Ναι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ε, ίδια σχόλια με τον εισηγητή έχω. Νομίζω ότι όντως είναι σαφές να ορίσουμε ποια θα είναι αυτά τα επόμενα βήματα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν αυτό το κείμενο από τον εισηγητή, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία και πρέπει να δούμε ποια θα είναι όντω η πραγματική συμβολή αυτού του εγγράφου. Η Κομισιόν κάνει κάποιες ε, προτάσεις σε διάφορους τομείς ε, και Ακούσαμε βέβαια και χτες κάποια στοιχεία έτσι, ακροθυγός για το cloud computing. Έχουμε τώρα τη νέα οδηγία για τα στατιστικά στοιχεία, για τα δεδομένα. Αν θέλουμε να επηρεάσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, προφανώς πρέπει να δώσουμε κι εμείς ε, κάτι. Να έχουμε δηλαδή ένα γραπτό πράγμα, κάτι απτό στα χέρια μας για να μπορούμε να το συζητήσουμε. Ε, φαντάζομαι ότι μέχρι, την, μέχρι το Γενάρη θα έχετε την υποστήριξη όλων των ομάδων. Επίσης το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δείτε γύρω μας τι γίνεται με τις τράπεζες και τις ε, ε, δαπάνες που έχουν. Τα θέματα ασφάλειας, ε, όλα όσα γίνονται γίνονται πια μέσω του ίντερνετ και εγώ έχω δέκα ανθρώπους που έρχονται και μου ζητάνε το, το password μου γιατί κάτι συμβαίνει και όλο λαμβάνω mail που λένε στείλτε μας το, το password. Κάποιοι δυστυχώς υποκύπτουν και το, και το δίνουν. Αλλά μιλούμε για τεράστια απάτη ε, μέσω του κυβερνοχώρου και αυτό το θέμα πρέπει να το θίξουμε. Για τη δική μου τη χώρα, ας πούμε, υπάρχει μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα, τους προσωπικούς λογαριασμούς, τους κωδικούς της κυβέρνησης. Και μπήκανε hackers σε αυτή την εταιρεία και όλα προφανώς κατέρευσαν. Οπότε θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή, από την 1η πρώτη του 12, γιατί το σύστημα αυτό τελικά απεδείχθη διάτρητο Οπότε, Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει καθημερινά και πρέπει να το σκεφτούμε. Πρέπει να δούμε και ποιε είναι οι οικονομικέ επιπτώσει όλων αυτών. Λοιπόν, ακούσαμε και από την Κομισιόν ε, χτε, από την Επίτροπο Κρούση, ότι θα υπάρξει ένα ε, πακέτο για την προστασία των δεδομένων με διάφορα άλλα στοιχεία. Βεβαίω θέλουμε να προχωρήσουμε, βεβαίω θέλουμε να υπάρξει πρόοδο. Εγώ απλώ απαντώ σε αυτά που ακούστηκαν από τον εισηγητή. Ε, Όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και βεβαίως όλοι ενδιαφερόμαστε να υπάρξει πρόοδος. Και βεβαίως έχουν γίνει ήδη πολλά, πρέπει να βασιστούμε σε αυτά. Η συζήτηση θα συνεχιστεί με την έκθεση Chichester στις αρχές του επόμενου έτους. Οπότε, και πάλι λέω, ε, συμφωνώ με αυτά που λέει ο εισηγητής, θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και Ευχαριστώ να τον βοηθήσουμε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, να ευχαριστήσω τους όσους πήραν το λόγο. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν εδώ που να θέλει το λόγο. Μάλλον εμείς φταίμε γιατί ε, πάμε πολύ γρήγορα σήμερα. Ε, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε το σημείο αυτό. Θα τα ξανασυζητήσουμε την επόμενη φορά. Πάμε στο σημείο 16. Ενημέρωση εκ μέρου ειδική αντιπροσωπεία του ΕΚ στην 6η συνάντηση Forum 2011 για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου 27-30 Σεπτεμβρίου στο Ναϊρόμπι. Εγώ δεν ήμουν παρόν. Οι συνάδελφοι που ήταν εδώ επίση δεν ήταν παρόντε και θέλαμε τόσο πολύ να ακούσουμε κάτι σήμερα και σήμερα δεν είναι κανένα εδώ που να πήγε στο Ναϊρόμπι. Η Πίλαρ Καστίγιο ήθελε να πάρει το λόγο και κάποιος μου είπε ότι έρχεται. Η κυρία δηλαδή μου είπε, η γραμματε... το μέλος γραμματείας μου είπε ότι έρχεται. Οπότε το θέμα είναι από πού έρχεται. Αν έρχεται από μακριά, α, μάλλον ήταν πολύ μικρός, ο, πολύ σύντομος ο δρόμος, από πολύ κοντά ερχόταν η συνάδελφος. Τέλεια. Κερδίζεις το βραβείο. Έχεις χρόνο ρεκόρ και δεν έχουμε και λουλούδια να σου δώσουμε. You can just start if you want. Αν θέλεις μπορείς να, να μας πεις δύο πράγματα, γιατί έχουμε τρεις ολόκληρους συναδέλφους που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για αυτό που έγινε στο Ναϊρόμπι. Α, υπάρχουν και γραπτές πληροφορίες, α, συνάδελφοι. Γι' αυτό δεν είναι εδώ οι υπόλοιποι που ήταν στο Ναϊρόμπι, γιατί τα έχουν διαβάσει τα κείμενα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ισπανικά για να τα πω ακόμη πιο γρήγορα. Όπως ξέρετε, από τις 26 έως τις 27, όχι, τις 27 συγγνώμη, ως 30 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα η, η έκτη συνάντηση Forum 2011 η διακυβέρνηση του διαδικτύου. Ήταν ένα φόρουμ το οποίο οργανώθηκε για πρώτη φορά στην Τίνιδα το 2005 και κάθε χρόνο γίνεται και σε διαφορετικό μέρος. Είναι περιπλανόμενο φόρουμ. Αυτό είναι ένα φόρουμ το οποίο οργάνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη και έχει παγκόσμιες διαστάσεις προφανώς και εκεί συμμετέχουν όλες οι περιοχές του πλανήτη μας. Φέτος η συνάντηση έγινε στο Ναϊρόμπι, πήγε μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, τρία μέλη του Κοινοβουλίου, μεταξύ αυτών και εγώ, ήμουν υπεύθυνη της αντιπροσωπείας και επίσης είχαμε και μια ευρύτερη εκπροσώπηση από την ε, Κομισιό. Η Νέλη Κρούς, η Επίτροπος, ήταν η επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κομισιό και συμμετείχε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες του φόρουμου και ήρθε και σε επαφή και με, την, με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης του Ναϊρόμπι, της Κένιας. Τα πιο σημαντικά θέματα, αυτά που ενδιαφέρουν το κοινοβούλιο μας δηλαδή, αφορούσαν το cloud computing. Αυτό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης. Επίσης η Κομισιό οργάνωσε ένα εργαστήριο για αυτό το θέμα και, σε, και όσον αφορά τις, ε, κυβερνητικές, τις υπηρεσίες, τον δημόσιο χώρο δηλαδή, Επίσης ε, οργανώθηκαν και άλλα ατελιέ σε συνεργασία ε, μεταξύ Αμερικανών, Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών εταιριών. Επίσης εργαστήρια για την προστασία των παιδιών και εκεί συμμετείχαμε όλοι μας. Το πιο σημαντικό από όλα είναι, τα, είναι το εξής κατά την άποψή μου. Το φόρουμ στο φόρουμ αυτό συμμετέχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τον τομέα, δηλαδή ε, επιχειρήσεις, ε, επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις καταναλωτών, κυβερνήσεις ε, κτλ. Δηλαδή συμμετέχουν πάρα πολύ και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ελέγχει τα όσα γίνονται είναι ένα φόρουμ όπου συζητώνται θέματα, δεν λαμβάνονται αποφάσεις ε, ε, σε νομοθετικό, σε κανονιστικό επίπεδο. Σαν φόρουμ συζήτησης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Γίνονται ανταλλαγές απόψεων, εκφράζονται όλες οι απόψεις Πρέπει να σας πω όμως το εξής. Η, επιτυχία αυτού του φόρουμ οδήγησε σε κάποιες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να αποκτήσει ένα πιο διακυβερνητικό χαρακτήρα. Και τελικά είναι οι κυβερνήσεις που εξασφαλίζουν την διαχείριση του φόρουμ. Δηλαδή η κυβέρνηση καθορίζει το πρόγραμμα και την συμμετοχή στο φόρουμ. Η Κίνα και η Ινδία ανέλαβαν κάποιες πρωτοβουλίες, το ίδιο και η Βραζιλία, όπως επίσης και κάποιες άλλες χώρες. Λοιπόν, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες έτσι ώστε το φόρουμ αυτό να μπορεί να λαμβάνει και αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά όμως υπήρχε το blog, το blog των Ευρωπαίων και των Αμερικανών που ήθελαν να το σταματήσουν αυτόν. Και η κυρία Κρούς και εμείς σαν βουλευτές επιμείναμε ε, ότι το φόρουμ αυτό πρέπει να διατηρήσει τον ε, ανοιχτό του χαρακτήρα. Γιατί και εκεί έγκυται και η χρησιμότητά του. Διότι αλλιώς δεν θα ήταν ένας τόπος συνάντησης, δεν θα είχε τον ίδιο χαρακτήρα, δεν θα, είχε την ίδια, δεν θα προσέφερε τις ίδιες δυνατότητε. Ήταν παρόν και ο Βρετανός Υπουργός Τηλεπικοινωνιών και συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις και είπε ότι δεν θα έπρεπε το φόρουμ αυτό να αποτελέσει ένα διακυβερνητικό εργαλείο. Υπογράμμισε ότι θα πρέπει να παραμείνει ο ανοιχτό χαρακτήρα του φόρουμ. Και αυτό. Αυτή ήταν η γενικότερη θέση, όπω σα είπα, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Λοιπόν, το θέμα θα ζητηθεί στα Ηνωμένα Έθνη και εκεί τα Κίνα, η Κίνα ίσως να ζητήσει να εγκριθεί ένα ψήφισμα ε, όπου θα παρουσιάζεται η θέση της οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλες δυτικές χώρες ε, έχουν ε, διαμορφώσει συγκεκριμένη θέση. Ε, επίσης θα πρέπει να σας πω και για τις επαφές που είχαμε με την κυβέρνηση της Κένιας. Η Κένια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα. Αναπτύσσεται η Κένια έχει σημαντική οικονομική ανάπτυξη. Είναι επικεφαλής, αν θέλετε, των ε, χωρών της ε, Ανατολικής Αφρικής. Και προφανώς χρειάζεται τεχνολογία, εφαρμόζει ε, την πληροφορική, την, την τεχνολογία της, των τηλεπικοινωνιών κτλ επισκεφθήκαμε ένα σχολείο όπου φοιτούν 2.000 παιδιά. Με την κυρία Κρούς. Το σχολείο αυτό βρίσκεται σε μια φτωχιά γειτονιά θα τη χαρακτήριζα του Ναϊρόμπι. Όμως το σχολείο αυτό είχε τονίσει μία πτυχή της εκπαίδευσης που ήταν η τεχνολογία της προφορικής και της επικοινωνίας. Πραγματικά τα επιτεύγματά τους ήταν εντυπωσιακά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βρίσκουμε, το συναντάμε συχνά στην Κένια. Ο διευθυντής του σχολείου εξέφρασε την επιθυμία το φόρουμ αυτό να παίξει, να παίξει ένα κάποιο σημαντικό ρόλο. Ούτως ή άλλως η προετοιμασία του κράτησε ένα χρόνο σχεδόν. Το Δεκέμβριο θα γίνει και ένα debriefing με την, με την και επαναλαμβάνω ότι θέλουμε να παραμείνει ο ανεξάρτητος και ανοιχτός χαρακτήρας του φόρουμ αυτού. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά σαν και αυτό το φόρουμ σήμερα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Βέβερα έχει ένα ερώτημα. Euh, Ευχαριστώ για αυτήν την παρουσίαση που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έχετε δίκιο στα συμπεράσματά σας για να διατηρήσει αυτό το φόρουμ το χαρακτήρα της ανοιχτής συνέλευσης, συγκέντρωσης για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων. Θα ήθελα όμως ως προς το θέμα αυτό να σας θέσω μια ερώτηση. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον τομέα ακριβώς των νέων τεχνολογιών είναι αυτό που ονομάζουμε ε, το χάσμα το ψηφιακό που έρχεται και προστίθεται σε χάσμα οικονομικό και σε χάσμα κοινωνικό. Γι' αυτό ε, με ενδιαφέραν αυτά που είπατε σχετικά με τη γένεια και την, το παράδειγμα αυτής της σχολής, σε αυτό το φόρουμ. Γίνονται προτάσεις ε, για να αποφύγουμε την διεύρυνση αυτού του ψηφιακού χάσματος, ούτως ώστε οι τεχνολογίες αυτές ε, να ε, αναπτυχθούν, για να αναπτυχθούν χρειάζονται επενδύσεις σημαντικές και για την πρόσβαση στις τεχνολογίες αυτές απαιτούνται ε, μεγάλες επενδύσεις ε, στις χώρες, στις ακτές υπάρχουν αυτές οι επενδύσεις αλλά όλοι μένουμε στην ενδοχώρα δεν υπάρχουν τέτοιες επενδύσεις ασχολήθηκε το φόρουμ αυτό το θέμα και έχουν υποβληθεί προτάσεις ούτως ώστε ε, να μην διευρυνθεί και να μην παγιωθεί αυτό το χάσμα, να μην εδρεωθεί. Ευχαριστώ. Απλώς μια ερώτηση που θα ήθελα ε, να θέσω, διότι νομίζω ότι το θέμα δεν συζητήθηκε στο φόρουμ, αλλά θα πρέπει και η Επιτροπή μας να ασχοληθεί. Είναι το νέο πρωτόκολλο, διεθνές πρωτόκολλο. Ίσως ασχοληθήκατε με το σημείο αυτό το, ε, το ε, πρωτόκολλο που υπάρχει για το διαδίκτυο έχει εξαντληθεί, έχει λήξει, υπάρχει νέο σχέδιο και ίσως κάποια στιγμή θα ε, θα, δεν θα έχουμε πλέον ε, διευθύνσεις ε, διαδικτύου και το πέρασμα στο νέο πρωτόκολλο απαιτεί προσπάθειες που δεν γίνονται μόνο πάνω σε εμπορική βάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να μελετά κάποια στρατηγική, ένα κείμενο για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Κομισιό, ούτως ώστε να βελτιωθεί το κείμενο αυτό. Βλέπω ότι χρησιμοποιήσατε την, ε, συζητήσατε το cloud ε, computing από ε, δημόσιους οργανισμούς. Εδώ δεν γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι έγινε. Πίλα, please, yeah. Sí, eh, vamos a ver. En relación a la, a la Λοιπόν, σε σχέση με την πρώτη παρατήρηση, es, eh, για, τα ε, ε, ψηφιακά τιμολόγια κτλ. Η συζήτηση είναι ανοιχτή ούτω ή άλλω για το πώ βλέπουμε το θέμα από κοινωνική και οικονομική πλευρά. Και το συζητάμε προφανώ και, ε, και στο φόρουμ. Εκτός όμως από μια απλή, ένα απλό κατάλογο ενεργειών που θα πρέπει να αναλυθούν, είναι και θέμα γενικών προσανατολισμών. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και όχι μόνο απέναντι στις χώρες μας, Αυτά τα συζητάμε όταν ε, ασχολούμεθα με την, υψηλή, υψηλή, με την διαβίβαση στοιχείων υψηλής ροής και τα λοιπά, με υψηλή ροή Και, τα λοιπά. και να ξέρουμε τώρα όμως βέβαια και από ποια σκοπιά μιλάμε, από την Κομισιό, από το Κοινοβούλιο, από την κυβέρνηση. Από πλευράς του ΕΛΚ είναι ένα από τα θέματα τα οποία ετέθησαν όταν συζητήσαμε με τους βουλευτένιες και με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Γερμανία, από τη Γαλλία νομίζω και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούστηκαν κάποια ερωτήματα και ένα από τα ερωτήματα αυτά ήταν το επόμενο, στο επόμενο φόρουμ για τη διακυβέρνηση να προβλέπεται ένας χώρος για τους ε, εκπροσώπους των διαφόρων κοινοβουλίων. Και με την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκεί να συζητηθούν τα ε, ερωτήματα τα οποία και εσείς θέσατε. Βέβαια, έχουν αναλυφθεί πολλές πρωτοβουλίες, υπάρχουν πολλά προγράμματα. Συμμετείχαμε στην παρουσίαση ενός προβλα... προγράμματος για την ε, επαναχρησιμοποίηση της τεχνολογίας. Μία εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα ασχολείται με αυτή την ανακύκλωση των, του τεχνολογικού εξοπλισμού και πολλά από αυτά που είχαμε χρησιμοποιήσει εμείς ήταν αποτέλεσμα ανακύκλωσης. Τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων προσόντων που αφορούν την τεχνολογία. Τώρα σε σχέση με αυτά που είπε ο συνάδελφος, για το ICAN και το πρωτόκολλο, να σας πω, συμμετείχαμε σε μία συνάντηση. Tenemos ε, muy poco que hacer porque desde el punto de vista de ε, se Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τις ερωτήσεις μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει και αρμοδιότητες. Η ΑΕΚΑΝ είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία ασχολείται με την διαχείριση και η οποία έχει συνάψει μια συμφωνία με την ε, κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ο τρόπος λειτουργίας του ICAN όσον αφορά την διαφάνεια, τη συμβατότητα, τα μέλη του, ε, του Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να διευκρινιστούν στο Συμβούλιο, στο Συμβόλιο, συγγνώμη, ανάμεσα σε μια κυβέρνηση και την επιχείρηση αυτή. και είναι θέμα προσέγγισης κιόλας και αντιμετώπισης πιστεύω. Ούτως ή άλλως είναι και θέμα λίγο πολύ μονοπωλίου, δεν είναι ανοιχτή η αγορά. Και εφόσον υπάρχει μόνο αυτή η επιχείρηση, αυτή η επιχείρηση μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά, η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι δεν λειτουργούμε σε μια ανοιχτή αγορά, με μια αγορά με ελεύθερο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά όσον αφορά ε, την διαφάνεια και την συμβατότητα που σας είπαμε και τη συμμόρφωση. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες ούτως ή άλλως η ευθύνη της ε, επιχείρησης αυτής ε, είναι ακόμα μεγαλύτερη και το ξέρει αυτή η, η εταιρεία. Ξέρει ποια είναι η θέση της ε, στο, στο, χώρο, στο του ίντερνετ, ο οποίος δεν έχει και όρια ούτως ή άλλως. Εμείς αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε είναι να υπογραμμίσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν Λοιπόν, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση που είχαμε με την Ικάνο. Και ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε. Δεν ε, θίξαμε το τεχνικό αυτό ζήτημα το οποίο εσείς αναφέρατε, γιατί δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο εξάλλου. Για την επόμενη συνάντηση θα ήθελα να ζητήσω, αν γίνεται, να συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής, διότι πιστεύω ότι τότε θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι και οι μελλοντικές μας ενέργειες. Αυτά. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, όλοι την έχουμε την ε, έκθεση. Έχουμε μάλιστα και ένα, μια, έτσι, ένα κείμενο με πολλές φωτογραφίες ε, από το Ναϊρόμπι. Η ε, γραμματεία μου, λένε, μου λέει να, αν θέλουν κάποιοι να αλλάξουν το κείμενο αυτό που ήταν στο Ναϊρόμπι, θα πάει, έχετε μια εβδομάδα. Αλλιώ θα πάει στο, να τυπωθεί και θα δημοσιευθεί. Οπότε κλείνουμε το σημείο αυτό. Οπότε, όχι δεν κλείνουμε ακόμα. Ε, πρέπει να ε, ευχαριστήσουμε τη Γραμματεία, Πρόεδρε, γιατί ήταν εξαιρετική. Η Λίνα ήταν μαζί μας και πάρεμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από την ε, Γραμματεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ. Το χαίρεται και η Γραμματεία, βεβαίως και εμείς. Ευχαριστούμε μέσω ημών τη Γραμματεία για την εργασία της. Οπότε κλείνουμε τη συνεδρίαση. Καλό μεσημέρι εύχεται ο Πρόεδρος και στους διερμηνείς. Οπότε έχουμε όλοι μεγαλύτερο, α, μεγαλύτερο διάλειμμα και τα λέμε το μεσημέρι.